Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δυστυχώς η ώρα να αρχίσουμε αν και λείπουν οι περισσότεροι. Αλλά έχουμε ήδη καθυστερήσει 12 ολόκληρα λεπτά. Και μετά θα μιλήσουμε για το σημείο 27. Uh, και θα δούμε την, ε, το σχέδιο εκθέσεις Uh, για τα καζεϊνούχα. Σύμφωνα με την οδηγία 83 κάθετος 317 κάθετος ΕΟΚ. Και θα δώσω στον εαυτό μου το λόγο ως εισηγητή. Ως εισηγητή. Τον Μάρτιο του 2014 δημοσιεύθηκε η πρόταση οδηγίας για τη γυθνίαση ε, των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την καζεΐνη και τα καζεϊνούχα. Ε, προτείνεται να πάψει να ισχύει η οδηγία του 2005 η σχετική με τις ε, γαλακτοπρωτεΐνες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτον, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των εκτελεστικών πράξεων και μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων, δεύτερον για να προσαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις της εξελίξεις της οδηγίας για τα τρόφιμα και τρίτον για να προσαρμοστεί και να ενημερωθούν οι τα προαπαιτούμενα χρήση των καζεϊνούχων στον λεγόμενο κώδικα τροφίμων, το κόντεξ αλιμεντάρις. Ε, ορίζεται στο 12% το ανώτατο ποσοστό υγρασίας που ήταν 10% στην προηγούμενη ρύθμιση. Το λίπος ε, μπορεί να φτάσει το 2% της καζεΐνης ενώ προεβλέπεται στην προηγούμενη ρύθμιση 4% για να υπάρξει γρήγορη προσαρμογή λοιπόν στα σημεία 1 και 3 στους κανόνες δηλαδή οι οποίοι εφαρμόζονται ε, στην, στην διατροφική καζεΐνη και ε, στην χρήση για τεχνολογικούς λόγους όπως επίσης και για την προσαρμογή στο νέο ε, διεθνές πλαίσιο προτείνεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η υιοθέτηση κατεξουσιοδότηση πράξεων τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ε, ε, στόχο τον τελικό καταναλωτή αλλά την βιομηχανία και γι' αυτό είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι στην διατροφική αλυσίδα να έχουν ε, τις απαιτούμενες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργογόνα. Η συμπερίληψη λοιπόν στην ετικετιστασία, στην σήμανση των καζεϊνούχων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση θα πρέπει να αναφέρεται και αυτό στο άρθρο 5. Τα προϊόντα αυτά αν δεν περιγράφουν στην συσκευασία τους το τι είναι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη χρήση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την προετοιμασία και προπαρασκευή τροφίμων. Πρέπει να αναφέρονται λοιπόν συγκεκριμένα οι αλλεργίες, αναφυλαξίες κτλ που μπορεί να προκληθούν από το συγκεκριμένο προϊόν. Ε, σχετικά τώρα με την προσαρμογή στον κόντεξ αλιμεντάριος, του οποίου τη σημασία αναγνωρίζουμε, είναι κάτι που θα δώσει εγγύηση ισότιμης μεταχείρισης σε όλους τους εμπλεκομένους στην αγορά. Προτείνονται κάποιες τεχνικές προσαρμοστικές διατάξεις Αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 5, στο σημείο 2 και στην τροπολογία 2, σημείο 7. Έτσι λοιπόν η κατεξουσιοδότηση πράξης ε, δεν ε, θα πρέπει να έχουν ισχύ βέβαια για ε, μία περίοδο αόριστη, αλλά για μία πενταετία, όπως ακριβώς έχει ισχύσει και για άλλες νομοθετικές προτάσεις του πεδίου ενδιαφέροντός μας. Τώρα η οδηγία αυτή βρίσκεται υπό εξέταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η θέση σε ισχύ της λειτουργίας ε, για δύο μήνες μετά την ψήφισή της είναι ε, φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική. Αλλά η πρόταση της Επιτροπής για τον μήνα Μάρτιο είναι υπερβολικά φιλόδοξη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό επιστρέφω και ξαναγίνομαι πρόεδρος και θα δώσω το λόγο τώρα στους σκιώδης εισηγητές. Θα ξεκινήσω με την συνάδελφο Μελιόρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και ως πρόεδρο αλλά και ως εισηγητή. Σωστά είπατε ότι είναι τεχνική αυτή η οδηγία για την οποία σήμερα μιλούμε Παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεστε. Oh. Είπατε κύριε Σιγητά ότι είναι ουσιαστικά τεχνική αυτή η οδηγία το 1983 ήδη που θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη νέα πρόταση και δεν αφορά τους τελικούς ε, καταναλωτές αλλά τους παραγωγούς ε, τις εταιρείε που χρησιμοποιούν καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα. Βέβαια, ε, είπατε και εσείς ο ίδιος ότι είναι σημαντική η πληροφόρηση και η ενημέρωση για να ε, ξέρουμε στη συνέχεια και τι μπαίνει στα γαλακτοκομικά προϊόντα και αυτό να γνωρίζουν οι καταναλωτές. Ιδιαίτερα οι αλλεργικοί καταναλωτές ε, γιατί αναφέρονται τα αλλεργιογόνα. Υποστηρίζουμε την τροπολογία ε, μάλλον να το πω αλλιώς, την τροποποίηση, τον τρόπο με τον οποίο εσείς αλλάξατε την έκθεση. Auch alle anderen... ε, όλες τις άλλες ε, προτάσεις σας ε, τις υποστηρίζουμε φυσικά κι εμείς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρότασή σας και ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα. Ωστόσο έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η οδηγία του 83 που θα πρέπει να αντικατασταθεί έχει ένα άρθρο 7 εδάφιο 1 που αναφέρει μια ασφαλιστική δικλίδα, μια ρήτρα ασφαλείας ας πούμε, όταν πρόκειται για κίνδυνος για, τη, για κινδύνους για δημόσια υγεία υπάρχουν δυνατότητες για τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν τη χρήση στην επικράτειά τους. Αυτή η ρήτρα έχει πλέον εξαφανιστεί και ρωτώ για ποιο λόγο. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά μου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η παραγωγή κασεΐνης. 15.000 τόνους παραγάγαμε πέρυσι που αντιπροσωπεύουν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι σημαντική και για τα γαλακτοκομικά γενικότερα. Επίσης χαίρομαι για την ενημέρωση αυτή γιατί η προηγούμενη νομοθεσία είναι από το 1993 και καλό είναι να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν καινοτομίε. Ας πούμε το ανακάτεμα του γάλακτος με μεμβράνες και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι νέες τύπου τεχνολογίες και τεχνικές να λαμβάνονται υπόψη. Γι' αυτό συγχαίρω τον εισηγητή που τα είπε πολύ καλά και θα τον υποστηρίξω, θα τον υποστηρίξω. Μία μόνο αντιρρησούλα και τροπολογία θα καταθέσω για να ευθυγραμμιστεί τελείως με τα πρότυπα του ΒΟΕ και του ΦΑΟ. Εγώ σας ευχαριστώ. Άμα θέλω μιλάω και 30 λεπτά, ε, αλλά ίσως και λιγότερο. Λοιπόν, είναι τεχνικό το θέμα και αν και είναι σημαντικό, δεν θα καταθέσουμε καμία ντροπολογία γιατί δοχόμαστε και καταλαβαίνουμε αυτά που είπε ο εισηγητής. Χαρείτε όσο μπορείτε. Και πράγματι η Κομισιόν τώρα προσπαθεί με την προσθήκη να κινηθεί προς κατεξουσιοδότηση πράξη, αν και όταν πρόκειται για θέματα τύπου TTIP ε, δεν μας αρέσει πάντοτε, αλλά σε αυτή την περίπτωση φαίνεται λογικό για να διευκολυνθούν οι αλλαγές. Ακολουθούμε και σε αυτό λοιπόν τον εισηγητή. Συγχαρητήρια και τελειώνω την 25 λεπτή ομιλία μου έτσι. Φέτος, αυτό το απόγευμα έχουμε χρόνο, αλλά δεν πειράζει, ωφελήθηκες. Τώρα θα δώσω το λόγο για να δω ποιος κανείς, καμία, στην Κομισιόν για να απαντήσει στο μοναδικό ερώτημα που έθεσε η κυρία Μελιόρ. Ορίστε. Thank you, Mr. Chairman, and Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και το λόγο για αυτό το τεχνικό μεν πλην σημαντικό θέμα. Δεν ήθιστε εδώ στην Επιτροπή σας να έρχεται κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, της Γεωργίας δηλαδή και όχι της ε, Δημόσιας Υγείας, σαν πρώην και νυν σάντε. Εμείς κάναμε αυτή την πρόταση λοιπόν από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε το γαλακτοκομικό τομέα, ε, να είμαστε ε, στους ίδιους κανόνες ε, παιχνιδιού με τους ανταγωνιστές μας. Τόνισε μόλις ένας ευρωβουλευτής ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την γαλακτοπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την απασχόληση, για την ανάπτυξη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χαρά βλέπουμε ότι υποστηρίζετε την πρωτοβουλία μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το άρθρο 7, εδάφιο 1 της οδηγίας του 83, όπως είπε η κυρία Βουλευτής, εκεί υπήρχε μία διακριτική ευκαιρία για τα κράτη-μέλη να επεμβαίνουν σε περίπτωση κινδύνου δεν χρειάζεται πλέον αυτή η ρήτρα ή αυτό το άρθρο και η πρόνοια στη συγκεκριμένη πρόταση, διότι έχει ενσωματωθεί πλήρως στις συνθήκες και στις γενικές αρχές ε, για το δίκαιο που διέπει τα τρόφιμα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβουμε την ιδιαίτερη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη όταν ε, υπάρχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία να μπορούν να προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες. Γι' αυτό απλούστατα δεν το έχουμε επαναλάβει. Τότε το 1983 που ε, εγκρίθηκε αυτή η οδηγία ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Τώρα έχει γίνει ε, γενικός κανόνας αυτός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. δύο πολύ μικρά τεχνικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε, για τις τροπολογίες που προτείνατε εσείς, κύριε Σιγητά μου. Ίσως να σφάλω, διορθώστε με παρακαλώ, στην τροπολογία 2 που αναφέρεστε στην αιτιολογική σκέψη 7, η αιτιολόγησή σας πολύ σωστά επικεντρώνεται στο εξής γεγονός. Ε, τεχνολογικά ε, έκδοχα, δεν είναι ακριβώς έκδοχα, είναι προσθετικές ουσίες ε, και είναι είτε οξέα είτε αλκαλικά. Σωστό είναι αυτό. Στην τροπολογία σας χρησιμοποιείτε τον όρο processing aids που είναι ουσίες που υποβοηθούν τη διαδικασία. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα αλλά η διατύπωση έχει σημασία. και υποσημείωση αυτή που κάνω. Στη δε τροπολογία υπό αριθμό 5 έχω μια παρατήρηση για να βεβαιωθούμε ότι εννοούμε το ίδιο ακριβώς και κατανοούμε ε, με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση και εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο και εμείς στην Επιτροπή. Τι εννοώ. Αν ε, κατάλαβα καλά, προτείνεται η ελάχιστη περιεκτικότητα στη γαλακτοπρωτεΐνη καζέινη να μην υπολογίζεται επί της ξηράς ουσίας, αλλά επί του συνολικού βάρους του προϊόντος. Δηλαδή 88% διατηρείται αυτό, αλλά αναφέρεται ε, με βάση ε, το βάρος του προϊόντος, αλλά έχει τη ξηρά ουσία. Ναι, αλλά έτσι νοθεύεται ο ανταγωνισμό απέναντι στους ανταγωνιστές μας. Και όπω είπε κάποιο βουλευτή προηγουμένω, ανέφερε κάποια στοιχεία για την γαλακτοπαραγωγή και για τις εξαγωγές και θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το στοιχείο. 50% των, ε, της καζεΐνης που παράγουμε το εξάγουμε. Δηλαδή είναι ένα υψηλής ποιότητας ε, προϊόν για το γαλακτοκομικό τομέα. Εισάγουμε ελάχιστες ποσότητες και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό όχι για ανθρώπινη κατανάλωση. Οπότε δεν υπάρχει απειλή από τις εισαγωγέ από τρίτες χώρες του ή πιν. Και θέλουμε πραγματικά να ε, ευθυγραμμιστεί ε, ο κλάδος στην Ευρώπη με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές. και θέλουμε να σας προτείνουμε να γίνει το υπολογισμός βάσει ξηράς ουσίας. Ε, πράγμα που αναφέρεται και στο κόντεξ αλιμεντάριου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ και για τις χρήσιμες προτάσεις σας. Να ενθυμίσετε το χρονοδιάγραμμα 3 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι και προβλέπεται η ψηφοφορία στις 23-24 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας. Περνάμε στο επόμενο σημείο τώρα της ημερήσιας διάταξης στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. Όπως γνωρίζετε η Επιτροπή Ήτρε είναι η υπεύθυνη επί της ουσίας και θα έχουμε μία συζήτηση πάνω σε αυτό. θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της η κυρία Κίλονεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε για τα θέματα της ενέργειας. Όταν συζητάμε για αυτό το θέμα, έχουμε να κάνουμε με μία ανάγκη όλων των κατοίκων της Ευρώπης. Πολύ συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένουμε εγγραφόμεθα σε ένα γενικό πλαίσιο. Μιλάμε δηλαδή για τις απειλές <clears throat> και την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας αλλά για τους πολίτες μας. Το θέμα είναι πιο συγκεκριμένο, να μπορεί να ζεσταίνει κανείς το σπίτι του, να έχει φως, να έχει μια αίσθηση ασφάλειας. Πρέπει φυσικά να μιλήσουμε και για τα στρατηγικά θέματα, πρέπει να μιλήσουμε και για την εξάρτηση και για το χρήμα και τις υποδομές. Πριν από οτιδήποτε άλλο όμως να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω πως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο συνάδελφός μας ο κύριος Σιλικιώτης το ανέφερε αυτό στα πλαίσια ε, των συζητήσεων της ΣΥΤΡΕ. Πρέπει να διασφαλίσουμε την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους πολίτες με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Και οι φτωχότεροι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Η έμβια η ενεργειακή δυστυχώς είναι κάτι που χτυπά το 20% των Ευρωπαίων ενώ οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν και τα πράγματα γίνονται πολύ περίπλοκα. Υπάρχουν και κάποιες ειδικέ καταστάσεις οι οποίες έχουν σχέση με τις κλιματολογικές αλλαγές. Εισαγωγές, εξαγωγές και όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχωρίζουμε από την καθημερινότητα των πολιτών. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο μας καθιστά ευάλωτους. Εισάγουμε πάνω το 50% της ενέργειας που χρειαζόμαστε και είμαστε εξαρτημένοι από το πετρέλαιο. Το κόστος για την κατανάλωση υγρών καυσίμων είναι ιδιαίτερα υψηλό σε καθημερινή βάση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ε, εξοικονομήσεις και στον τομέα αυτό και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το κέντρο των ανησυχιών μας. Απαιτείται να είμαστε ε, πολύ πιο αποτελεσματικοί στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας, να μειώσουμε τις εκπομπές Απαιτείται μια κοινή στρατηγική και αυτό είναι η απάντηση σε πάρα πολλές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα που συνδέονται με τις κλιματολογικές αλλαγές γενικά με ένα πακέτο για την αηφορία στην ενέργεια και τις καινοτόμες τεχνολογίες τις οποίες και αυτές θα πρέπει να αναπτύξουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να μας απασχολήσουν παράλληλα. Απαιτείται ανάληψη δράσης τώρα, δεν έχουμε χρόνο. Στόχος μας, μακροπρόθεσμα, είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ορυκτά καύσιμα το 2050 σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Ήδη από το 20 θα έχουμε μειώσει τη χρήση τους. Οφείλουμε να δράσουμε λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους επιγόντως. Ε, για τα κτίρια και για τις μεταφορές πολλά μένει να γίνουν. Τα αποτελέσματα θα τα πετύχουμε μόνο αν συνεργαστούμε ε, με τα κράτη-μέλη ε, με αγαστό τρόπο. Έτσι θα ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα δράσης και κάποια νομοθετικά κείμενα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να υπάρξει ανάκαμψη της έρευνας και να αναπτύξουμε τεχνολογίες που θα μας επιτρέψουν να αποκλίνουμε από την χρήση των ορυκτών καυσίμων. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν θα πρέπει να αγνοηθούν συνεπώς. Ήδη σήμερα υπάρχουν κάποιες λύσεις οι οποίες θα γίνουν πιο συγκεκριμένες και για την αποθήκευση της ενέργειας και η καινοτομία εδώ είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τους εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων για όλα αυτά και στο σχέδιό μου προσπάθησα να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες και τις ελπίδες του καθενός. Δεν θα υπάρξει βέβαια δυστυχώς από μια άποψη επανάσταση στον τομέα της ενέργειας, αλλά περιμένω με ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις τις οποίες θα κάνετε. Για να τελειώσω θα ήθελα να επανέλθω για μια ακόμη φορά στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Εγώ έρχομαι από τη Βόρεια Φιλανδία, από την περιοχή του Καϊνού ε, η φύση εκεί βρίσκεται στο κέντρο της ζωής μας και οι κάτοικοι της περιοχής έδιναν μάχες για να επιβιώσουν. Και αυτό το οποίο μάθαμε από αυτή τη μάχη είναι ότι ο καθένας θα πρέπει να προσέχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Γιατί αν δεν σκέφτεται το τι τον περιμένει αύριο τότε δεν θα έχουμε μέλλον. θα πρέπει να μπορούμε να διατηρούμε τις πατάτες στα σπίτια μας για να βγάλουμε το χειμώνα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε, να κυνηγούμε ε, άγρια ζώα για τροφή. Λοιπόν, όλα αυτά στα πλαίσια της ενεργειακής αποδοτικότητας, ε, αν τα πετύχουμε όλα αυτά, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα. Siksi Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι το βασικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλα τα, τις ομάδες για τη συνεργασία τους. Σας Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει κυρία Γκαντίνη. Να πω αμέσω στους συναδέλφους ότι για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, θα ήθελα να αντικαταστήσω τον συνάδελφο Μέλιο που μου ζήτησε να σας μεταφέρω ε, κάποια σημεία τα οποία μου έδωσε για τα οποία ε, η ίδια δεν μπορεί να είναι παρούσα. Την επόμενη φορά νομίζω ότι θα είναι πιο, ε, πιο πλήρης από εμένα. Καταρχάς, η ευημερία και η ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης εξαρτάονται από μια ουσιαστικά ασφαλή και πλούσια προμήθεια ενέργειας. Οι μηχανισμοί ενέργειας που υπάρχουν θα πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει προβλήματα διακοπής προμήθειας ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι εννοεί κανείς ε, με την συγκεκριμένη φράση. Έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις, αλλά έχοντας ακούσει και την εισαγωγή της κυρίας Κιλόνεν, είναι σαφές ότι εδώ είναι ένα μέτωπο στο οποίο θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα βήματα προς τα εμπρός. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τον συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών για να ενισχύσουμε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσει ε, ε, νόμους οι οποίοι να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Η ενεργειακή αγορά πρέπει να συμπληρωθεί, πρέπει να υπάρξει μια λειτουργική και ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας, πρέπει να αναπτυχθούν οι διασυνδέσεις θέτοντας τέλος στην απομόνωση κάποιων κρατών μελών που θα πρέπει να συνδεθούν με τα υπάρχοντα δίκτυα. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει την διασφάλιση της προμήθειας ενέργειας αλλά και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την αύξηση του ανταγωνισμού. Οι κατάλληλες ενεργειακές διασυνδέσεις και η ολοκλήρωση της αγοράς της εσωτερικής ενέργειας είναι οι δύο πυλώνες εξυγχρονισμού της ενέργειας στα κράτη-μέλη και αυτό μπορεί να γίνει με αποτελεσματικό τρόπο και σε επίπεδο κόστους, εξυπηρετώντας στόχους ευεργετικούς και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς. Πρέπει να προωθήσουμε την διαφοροποίηση των πηγών προέλευσης ε, των, ε, της ενέργειας και της οδούς ε, τις οποίες ακολουθούν. Το φυσικό αέριο φυσικά και ο ηλεκτρισμός εδώ είναι οι προτεραιότητές μας. Πρέπει να επενδύσουμε στην καθαρή ενέργεια ε, σαν παράδειγμα, παλήρια. Νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Οι επενδύσεις λοιπόν εδώ θα πρέπει να στραφούν και στις ανανεώσιμες πηγές και την ικανότητα της Ένωσης να τις εκμεταλλευτεί πλήρως. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος που είναι υπεύθυνη από της ουσίας την άλλη φορά θα σας τα πει καλύτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι θα επωφεληθώ της ευκαιρίας που μου δίνεται να μιλήσω στην Μαλτική. Και αρχίζω με τον, ε, ευχαριστώντας τον εισηγητή διότι οι περισσότερες προτάσεις την εισηγήτρια μας συμπεριλήφθηκαν. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι η βάση της ενεργειακής πολιτικής. Επειδή προέρχομαι από τη Μάλτα με μικρό και απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, ξέρω ότι δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε δεδομένη την ενεργειακή ασφάλεια και πιστεύω ότι η αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη και η ενεργειακή εμπιστοσύνη και ασφάλεια πρέπει να είναι πολύ βασικά στοιχεία της πολιτικής μας. Επίσης όλα δείχνουν ότι πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά γρήγορα. Αυτή τη στιγμή οι αλλαγές στην ενωσιακή αγορά βασίζονται στην έννοια της ε, ασφάλειας των πηγών και της μεταφοράς των αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δίνουν νέες ευκαιρίες να αυξήσουμε τη διαφοροποίηση της προμήθειάς μας από εκτός ένωσης και να βασιστούμε περισσότερο σε ενδογενή παραγωγή. Έχω πέντε σημεία. Πρώτον, για την διαφοροποίηση. Υπάρχει δυναμική για συνέργεια με χώρες από την Εγγύη Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Μεσόγειος γίνεται όλο και σημαντικότερη για αυτά τα πράγματα και ως προς τις υπάρχουσες πηγές και ως προς τις μελλοντικές και για αυτόν τον λόγο το σχέδιο ενός μεσογειακού κέντρου αερίου πρέπει να δημιουργηθεί. Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα καύσιμα για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το τωρινό επίπεδο εκπομπών αερίων με το πρασίνισμα του ηλεκτροδότησης και την ηλεκτροδότηση του μεταφορικού συστήματος ώστε να μειωθούν εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακος. Γι' αυτό βέβαια χρειάζονται και εναλλακτικά καύσιμα η χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου πρέπει να ενθαρρυνθεί για τα βαρέα οχήματα ακόμη και για τα πλοία. Τρίτον, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των ανανεωσίμων και της αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας χρησιμοποιώντας τα φωτοβολταϊκά και αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας με καινούριου σύγχρονους σύγχρονες γεννήτριες. Τέταρτον, θα ήθελα να γίνει περισσότερη έρευνα και καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, χρήση νέων τεχνολογιών, νέων μορφών ανανεωσίμων με πιο οικονομικό τρόπο. Από καλύτερη χρησιμοποίηση της ενεργείας των κυμάτων μέχρι τα φωτοβολταϊκά και τη χρησιμοποίηση φυκιών. Τέλος, αν και το σπουδαιότερο, πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι οι σταθερότερες βάσεις και προϋπόθεση για μια λειτουργούσα σωστά ενεργειακή αγορά. Βασικό στοιχείο γι' αυτό θα ήταν καμία χώρα μέλος να μην απομονώνεται από τα δίκτυα ηλεκτρικά και αερίου. Και επομένως και η μελλοντική αεριαγωγή που έχουν αρχίσει να σχεδιάζονται πρέπει να υλοποιηθούν γιατί αυτά είναι θέματα κοινού ευρωπαϊκού συνειφέροντος. Βυσνιέσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αντίθετα από τον συντάκτη. Νομίζω ότι τα προβλήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια δεν θα λυθούν μέσω κοινών δράσεων της Ένωσης. Αντίθετα, καμιά φορά η Ένωση περιορίζει τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων, των καταλληλότερων αποφάσεων από τα κράτη-μέλη, ιδίω ως προς τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι πηγές της χώρας, οι ενεργειακές πηγές και καμιά φορά το ότι να μπορεί η χώρα να αποφασίσει μόνη της είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει και το θέμα των υποδομών για την μεγιστοποίηση των πόρων σε εθνικό επίπεδο. Έχουν γίνει αναλύσεις και μελέτες για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αποθήκευση και νομίζω ότι στο μέλλον αυτό θα σήμαινε πολιτική όθηση της χρήσης του αερίου ιδίως με μακροπρόθεσμα συμβόλαια από τρίτες χώρες. Παρά τις αμφιβολίες μας λοιπόν για το κείμενο γνωρίζουμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αφορά ακόμη σύμφωνα με τη συνθήκη τα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για να καθορίσουν το ενεργειακό τους μείγμα. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακατεύεται παντού και μας το εμποδίζει. Σήμερα η κλιματολογική πολιτική δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη της την ποικιλομορφία που έχουν οι χώρες μέλη. Σε χώρες σαν τη δική μου την Πολωνία... δεν μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου χωρίς παράλληλα να αυξηθούν οι τιμές της ενέργειας. Αυτό θα έχει τελικές αρνητικές επιπτώσεις στα νοικοκυριά, στους χρήστες, στη βιομηχανία και όλα αυτά αντιβαίνουν στην έννοια την ίδια της ενεργειακής ασφάλειας που σημαίνει πρόσβαση στην ενέργεια μεν αλλά επίσης και λογικές τιμές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στόρβατς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Linux. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Κούλονεν για την εξαιρετική της γνωμοδότηση. Μεταξύ των όσων είπε, άκουσα ότι άκουσε λέει όλες τις πολιτικές ομάδες και σημείωσε τα σχόλια τους. Έχει δίκιο. Γιατί αυτά που ζητήσαμε εμείς οι φιλελεύθεροι τα έχει συμπεριλάβει. Συνεχίζω τώρα στα αγγλικά. Γνωμοδότηση είναι ε, και σε μία σελίδα είναι δύσκολο να χωρέσουν ε, όλες αυτές οι επιθυμίες για να φτιάξουμε ένα ευχολόγιο που να μην είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ε, τη της νομοδότησης ε, τα κατάφερε πολύ καλά και νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές τοπολογίες. Ξέρουμε φυσικά ότι έχουμε τεράστια εξάρτηση στην ε, Φιλανδία και στις χώρες της Βαλτικής από ορυκτά καύσιμα και πόσο μάλλον από την εισαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία. Ε, και αυτό έχει και μια ενδιαφέρουσα επιπλοκή. Ξέρετε ποιες είναι οι τεχνολογικές προδιαγραφές ε, στη Ρωσία και οι πολιτισμικές διαφορές που έχουμε. Στις πετρελοπηγές ε, και στις χώρους εξόριξης φυσικού αερίου είναι τεράστια η έκκληση ε, διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή όσο χαμηλότερη είναι η τεχνολογία και παλαιότερη τόσο περισσότερο διοξιδίου του άνθρακα εκλείεται. Άρα αν τους πιέσουμε να ε, ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον και για τις αξίες μας, θα βοηθήσουμε και τους ίδιους μας τους αυτούς. Αλλά θα πρέπει κάπως να διαφοροποιήσουμε και τις πηγές μας για να μειωθεί αυτή η εξάρτηση. Άρα χρειάζονται βιοκαύσιμα στο μέλλον και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις και την καινοτομία. Είναι σύντομη μεν η γνωμοδότηση, πλην ο δρόμο μακρύς ακόμα μπροστά μα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πεντησίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον, να εκφράσω το σκεπτικό μου και σε αυτά τα οποία είπε η συνάδελφος από τη σοσιαλιστική ομάδα η οποία αναφέρθηκε στα νέα από την Αφρικανική Ήπειρο στον τομέα της ενέργειας εδώ και λίγους μήνες. Τα πράγματα εξελίσσονταν συνεχώς λόγω των νέων μεθόδων εξαγωγής των υγρών καυσίμων με ε, μείωση στη συνέπεια της τιμής των μη συμβατικών καυσίμων όπως σαν παράδειγμα το φυσικό αέριο από σχιστολιθικές περιοχές. Βέβαια οι τεχνικές αυτές έχουν τεράστια ανάγκη ε, πετρελαίου και μία τιμή άνω των 85% το, το βαρέλι ε, πετρελαίου. Αυτός ο αγώνας λοιπόν ανάμεσα ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες, τη Ρωσία και την Σαουδική Αραβία ε, έχει αγνοήσει την φροντίδα για την υγεία των πολιτών ε, και την φροντίδα για το περιβάλλον. Βέβαια βραχυπρόθεσμα η εσωτερική παραγωγή θα έλυνε τα προβλήματα αλλά μακροπρόθεσμα όχι. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε ε, να υπάρξει μια απλήρης εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων και θα πρέπει η Επιτροπή μας να απελευθερωθεί από την εξάρτηση των, ε, των ορυκτών καυσίμων. Ευχαριστώ Μπάλτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αξιοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνετε. Τώρα που είμαστε και λιγότεροι συνάδελφοι και θα παρακαλούσα ή δυνατό να μιλήσω παραπάνω από 1,5 λεπτό. Αλλά απότε μου πει ο Πρόεδρος θα σταματήσω τι να κάνω. Πιστεύω ότι έχει σημασία και είναι και γεγονός ότι χρειαζόμαστε όλες τις πηγές ενέργειας. Όταν μιλούμε για ενεργειακή ασφάλεια, πάντα συζητούμε για υποδομές, για πρόσβαση στα δίκτυα, για ενεργειακές πηγές, αλλά πολύ σπάνια κοιτάμε τι σημαίνει η διανομή και ποιος είναι ο τελικός ε, στόχος. Να έχει ο κόσμος ενέργεια σε προσιτές τιμές η ομάδα των Πρασίνων είναι πάρα πολύ ριζοσπαστική στις απόψεις της. Και βέβαια όλοι ε, συμφωνούμε με αυτά που λέγουν οι Πράσινοι. Και βέβαια θεωρούμε όλοι ότι η ενέργεια είναι ένα κοινό αγαθό και θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι, να μην ε, έχουμε εξαρτήσει από το ρωσικό φυσικό αέριο προκειμένου. Όλα αυτά είναι ωραία και καλά να μην εξαρτώμαστε από διάφορους αγωγούς ε, διαμετακόμισης. Ωραία είναι όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση. Με την αιωλική ενέργεια και την ηλιακή. Δεν φτάνει για τις ανάγκες μας και για να είναι εξασφαλισμένος ο εφοδιασμός. Συμφωνούμε μεν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, αλλά και γι' αυτό χρειάζεται οικονομική υποστήριξη για να γίνει. Και όταν γίνεται λόγος για νέες τεχνολογίες, πάντα εμεί μιλούμε για ηλιακή, αιωλική και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να προσθέσω το εξή. Ήσασταν κι εσείς την προηγούμενη θητεία, εδώ θυμάστε το σχέδιο Desert Tech, που λέγαμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα της Ευρώπης ε, συλλέγοντας την ηλιακή ενέργεια στη Βόρεια Αφρική, στην έρημο και μεταφέροντας στην Ευρώπη την ενέργεια που θα παραγόταν εκεί. Τώρα όμως βλέπουμε ότι μετά την ε, Αραβική Άνοιξη να βάγισε αυτό το, πρόβλημα, το πρόγραμμα, συγγνώμη, Desert Tech. Αν προτιμούμε την αιωλική ενέργεια από την ηλιακή, έχει άλλο πρόβλημα, ότι δεν αποθηκεύεται η αιωλική ενέργεια. Οπότε δεν μας λύνει το πρόβλημά μας ούτε αυτή. Και είναι τελείως αστάθμητος παράγον. Για να έρθω τώρα όμως στην πυρηνική ενέργεια. Θέλουμε να μειώσουμε το, την εκπομπή διοξίδιου του άνθρακα. Όταν τα συζητάμε αυτά, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και την αμερικ... Ε, ενέργεια. Τέσσερις Αμερικανοί επιστήμονες συνέταξαν ανοιχτή επιστολή και τάχθησαν υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Και ένας από τους τέσσερις είπε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα η κλιματική αλλαγή, εξού και υποστηρίζω την πυρηνική ενέργεια και την ε, μεταξέλιξή της και την ανάπτυξή της. Και άλλοι όμως ε, επιστήμονες και ερευνητές εγνωσμένου κύρους ε, θεωρούν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ευκαιρία και διέξοδος. Αν θέλουμε λοιπόν να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, δεν επιτρέπεται να συζητούμε μόνο για την αιωλική και την ε, ηλιακή ενέργεια. Καλές είναι αυτές ανανεώσιμες να υποστηριχθούν και η έρευνα, αλλά χρειαζόμαστε και άλλες πηγές και θα πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα. Δεν φτάνουν αυτές οι πηγές αν δεν χρησιμοποιηθεί πυρηνική ενέργεια. Εγώ περίμενα να αντιδράσει ο κύριος Έκχαουτ πολύ έντονα σε αυτά που λέγω, αλλά έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Είμαι υπέρ μια στρατηγική ισόρροπης που θα ανταποκρίνεται και στα μελήματα των πρασίνων, αλλά δεν θα ε, ε, αρνείται την πραγματικότητα. Η κυρία Σχρέερ. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. 12 χρόνια στην Ολλανδία συζητούσαμε στο Κοινοβούλιο για την ενέργεια, όχι μόνο για την αιωλική ε, και την ηλιακή, γιατί μας φτάνει. Για να υπάρξει ενεργειακός ε, εφοδιασμός δεν φτάνουν οι αμυγός ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε και μια ενέργεια που να είναι αηφόρος και να είναι και προσιτή. Υπάρχουν ακόμα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και έχω επισκεφτεί και εγώ στο Χρόνιγκεν. Ε, πάνω από 3 δισεκατομμύρια κόστησε να φτιαχτεί το έργο. Είναι πάρα πολύ καθαρό, καμία σχέση με τα παλιά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Ένα δις ε, έχει έρθει ε, σε επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Καλό είναι να θέλουμε να αγοράσουμε καινούρια παπούτσια, αλλά για καλό και για κακό μην πετάξουμε τα παλιά πριν δούμε τα καινούρια. Κοινώς όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Ε, καλή η ενέργεια, η ανανεώσιμη ολική, ηλιακή. Ο κόσμος μπορεί να παράγει ε, ενέργεια με φωτοβολταϊκά για τον οικοκυριό του, για την γεωργική του εκμετάλλευση, αλλά το ε, πρόβλημα συνολικά δεν λύνεται Ο κύριος Γκρότε, και καλά, μην χαίρεστε και πολύ γρήγορα γιατί έφυγε ο Μπάσα Εκχάουτ, αλλά βάνω εγώ τώρα να μιλήσω σαν αυτόν. Ε, ωραίο είναι που συζητάμε αυτό το θέμα και τα κράτη-μέλη ε, είναι και παραμένουν αρμόδια για το ενεργειακό μείγμα. Δεν θα δοθεί εδώ αυτή η μάχη, ούτε πρόκειται να πείσω τους Πολωνούς ότι 85% άνθρακας δεν είναι καλό μείγμα στο δίκτυο διανομής, ε, ούτε πρόκειται να σας πείσω λέγοντας ότι έχουμε περίπου 95% της ενέργειας ε, στο δίκτυο ε, που δεν έχει καταρρεύσει ακόμα. Και θέλουν και οι Ολλανδοί να περάσουν υποθαλάσσιο καλώδιο για να παίρνουν φτηνό γερμανικό ρεύμα. Έρχομαι τώρα στην αιωλική ενέργεια. Αυτή θα πρέπει να είναι ε, για μας η στόχη. Εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους ε, και να υπολογίζουμε τι κοστίζει κάθε μορφή ενέργειας. Εδώ παραθέτουμε διάφορους επιστήμονες και διάφορα αριθμητικά στοιχεία ότι η πυρηνική ενέργεια 1,80 η κιλοβατόρα γιατί τα σκουπίδια κάπου πρέπει να τα ε, πετάξουμε τα ραδιενεργά απόβλητα δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε και έχουμε γενιές ολόκληρες ε, με ε, ρήπους, ε, πυρηνικά απόβλητα που πληρώνουν την κιλοβατόρα που έχει καταναλωθεί εδώ και αιώνες. Και μετά από 72 ώρες μπορούμε με 95% ασφάλεια να πούμε για την νεολική ενέργεια πόση ενέργεια παραμένει στο δίκτυο. Τα έχω συζητήσει αυτά τα θέματα και με τον κύριο Σεφσκοβιτς. Αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά ένα ευρωπαϊκό έργο χωρίς να τα ρίχνουμε ένα στον άλλον θα πρέπει να οργανώσουμε την ενεργειακή πολιτική. Και δεν θα πρέπει ο καθένας να έχει το δικό του δίκτυο ε, ανεξάρτητα και μεμονωμένα. Γιατί αυτό ε, δεν βοηθάει, ούτε οικονομίες κάνουμε, ούτε σταθερές τιμές έχουμε. Λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, να ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος τελικά, πόσο κοστίζει η κιλοβατόρα από την χή πηγή και αυτό που θέλω επίσης να υπογραμμίσω είναι κάτι που έχει να κάνει με το υγροποιημένο ε, φυσικό αέριο. Εκεί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, ε, ιδιαίτερα στην αυτιλία, ε, το είπε και η κυρία Ντάλη, και σε ό,τι αφορά τα ναυπηγεία είμαστε πρωτοπόροι και μπορεί η Ευρώπη να είναι στην αιχμή του δόρατος για αυτό το θέμα ιδιαίτερα ε, να έχουμε και συγκεκριμένες ε, ε, ζώνες, περιοχές, το έχουμε κάνει αυτό ε, στην Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μάχη υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που περνάνε ε, ε, πλοία με χαμηλές εκπομπές σε θείο. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και θέσεις στα ναυπηγεία που έχουμε χάσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Οπότε θα πρέπει να βρει εξέχουσα θέση και πρωταγωνιστικό ρόλο η πρόταση της κυρίας Ντάλη στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ Κύριε Δεμέσμακα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ενεργειακή ασφάλεια, τι εστί, για τους πολίτες είναι κάτι το προφανές. Αυτό το λέει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε πρόσβαση στην ενέργεια. Η ασφάλεια του ενεφοδιασμού είναι κάτι το οποίο επισκιάζεται από άλλες σκέψεις, αλλά ειλικρινά νομίζω έχει παρέλθει ο χρόνος. Παλαιότερα αυτό το θέμα ήταν μεγαλύτερη προτεραιότητα και η συζήτηση ήταν αφηρημένη. Να σας δώσω δύο παραδείγματα στη δική μου χώρα, το Βέλγιο δηλαδή. Ο κίνδυνος blackout είναι πραγματικός, διότι στο παρελθόν έχουν λάβει 180 αποφάσεις ενεργειακές και τους τελευταίους μήνες ε, έχουν συγκεκριμένα σχέδια για σταδιακή διακοπή του ρεύματος. Μα αυτά δεν είναι ε, πράγματα για την Ευρώπη, ούτε για τα νοικοκυριά, ούτε για την ε, οικονομία, ούτε για τη βιομηχανία, ούτε για τις επενδύσεις. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα ενεργειακό μείγμα. Δεύτερον, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Ουκρανία, τι μας έδειξαν. Ότι έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ε, ασφάλεια ανεφοδιασμού. Σήμερα είναι επίκαιρη συζήτηση με, από αλλαγή απόψεων που είχαμε την περασμένη Τρίτη με τον κύριο Σέσκοβιτ, που είπε ότι αυτό το θέμα απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τους στόχους ε, του 2030 και προς μια ανταγωνιστική οικονομία με λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Υποστηρίζουμε μια ενεργειακή πολιτική που να βασίζεται σε τρεις αρχές. Ε, να είναι ευθυνή η ενέργεια, να υπάρχει ενεφοδιασμός εξασφαλισμένος και να είναι βιώσιμη. Αυτά τα τρία. Η ενέργεια ε, έχει να κάνει και με την ενεργειακή απόδοση, δηλαδή να κάνουμε οικονομία στην ενέργεια. Και βέβαια παίζει ρόλο εκεί το θέμα της ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά πρέπει να υπάρχει πλήρης ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Είναι τεράστιες οι διαφορές. Υπάρχουν ε, μικρές χώρες πυκνοκατοικημένες όπως είναι ε, το Βέλγιο και η περιφέρεια μου, η Φλάνδρα, που είναι σχεδόν ένα τεράστιο αστικό κέντρο ολόκληρη, είναι διαφορετική η κατάσταση. Λοιπόν, χρειάζεται βιώσιμη λύση, εξασφαλισμένος ανεφοδιασμός και αηφορία. Θα πρέπει να ποντάρουμε στην ενεργειακή απόδοση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν μόνα τους και στο μέλλον ε, στα μέτρα τους το ενεργειακό μείγμα που θεωρούν ε, σκόπιμο. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Ντέμουρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή μας συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια είναι πολύ επίκαιρη. Πρώτον, αυτά που είδαμε στην Ουκρανία δείχνουν τη σημασία της, αλλά επίσης γίνεται συζήτηση και για την μελλοντική ενεργειακή ένωση και είναι σαφές ότι η σημερινή μας συζήτηση θα συνδυαστεί και με εκείνη. Δύο σχόλια. Πρώτον, Βλέπω συνένεση στη σημασία να παραμείνει ευρεία η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας και των διαφόρων πυλώνων αυτής. Δεύτερον, βεβαίως, εφού είμαστε στην Επιτροπή Περίφ, η σημασία των εναλλακτικών πηγών ενεργείας και των ανανεωσίμων. Για το πρώτο, η ευρεία έννοια της ενεργειακής ασφαλείας δηλαδή, είναι κάτι που το είπαμε και τον Μάιο στην ανακοίνωσή μας και αν τη δείτε θα διαπιστώσετε ότι εκτός από τα πολύ βραχυπρόθεσμα μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης που είχαμε πάρει η κύρια, το κύριο μέλημά μας ήταν τα μακροπρόθεσμα. Δεύτερον θέλουμε μία πλήρως λειτουργούσα εσωτερική αγορά Τρίτον, ήταν η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ενεργειακών τεχνολογιών για καλύτερη διασφάλιση των προμηθειών και πηγών μας και τέλος να μιλούμε με μια φωνή και εξωτερικά για την ενεργειακή πολιτική. προσβλέποντας πάντα στην Ενεργειακή Ένωση. Τώρα για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τις ανανεώσιμες, η Κομισιόν με κάτι που το δέχεται. Θέλουμε να θεωρούμε ότι η περισσότερη αποτελεσματικότητα έχει πολύ, πολλές προοπτικές και σημαίνει την φτηνότερη ενέργεια που μπορεί κανείς να έχει. Όπως είπατε, ο αντιπρόεδρος Εύκοβιτς πήγε στην Ήτρε και δήλωσε ρητά ότι η προσέγγιση μας για την ενεργειακή ασφάλεια και προσβλέποντας πάντα στην Ενεργειακή Ένωση είναι ανταγωνιστικό, βιώσιμο σύστημα και πολιτική και σε αυτό το πνεύμα θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια των εργασιών σας. Ευχαριστούμε. Και τώρα για την κατάληξη η συγγήτριά μας, κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσω προσπαθώντας να σας πείσω να αλλάξετε τη γνώμη σας. Κατανοώ τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν όλοι και σε εθνικό επίπεδο και ευρύτερα, αλλά είναι σαφές ότι η ενέργεια και η αποδοτικότητα της ενέργειας είναι κάτι στο οποίο όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε. Τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε δεν είναι υποχρεωτικά πολύ ακριβά και δεν απαιτούν υπεράθρωπες προσπάθειες. Συνεπώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από σήμερα να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες ε, να μας ικανοποιούν όλους. Είναι ένα πρώτο βήμα προς τα εμπρός. Είναι σαφές ότι όλα αυτά κοστίζουν βέβαια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και ο άνθρακας και το πετρέλαιο ε, με τον τρόπο τους απαιτούν εκατομμύρια ευρώ, ευρώ και κοστίζουν σε όλη την Ευρώπη υπέρογκα ποσά. Το θέμα είναι να στηρίξουμε τις εναλλακτικές λύσεις, ε, τις εναλλακτικές έρευνες και να μην συνεχίσουμε και εμένουμε ε, στη λογική του business as usual. Οι τοπικές παραγωγές ε, άνθρακα είναι ένας τρόπος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει βέβαια στην απασχόληση των κατοίκων μιας περιοχής αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει συνολικά να στραφούμε στην έξυπνη παραγωγή ενέργειας. Αυτή είναι η λύση. Εμείς σαν κοινοβούλιο πρέπει να το κάνουμε αυτό πρώτοι. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ενέργεια με ε, ε, ευέλικτο τρόπο και να διασφαλίσουμε την προμήθειά μας με καθαρό τρόπο. Η επιθυμία μου θα έλεγα είναι να μην μου στείλετε 800 τροπολογίες αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς θα το αποφασίσετε αυτό. Σας ευχαριστώ και εμείς ελπίζουμε να μην υπάρξουν τόσες πολλές τροπολογίες. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 3η Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΗ στις 18 ε, Μαρτίου. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα Πρόκειται για την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Ανάπτυξης για τα μαθήματα από την κρίση του έμπολα και πώς να βοηθήσουμε τις χώρες να αποτρέπουν τέτοιου είδους θέματα στο μέλλον. Ναι. Ξέρετε ότι η κρίση έμπολα ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν τον κόσμο τον τελευταίο χρόνο ναι. και το έχουμε επανειλημμένα πει στις συζητήσεις μας και στις συναντήσεις με τους προσκεκλημένους μας. Αποφάσισε η Επιτροπή Ανάπτυξης τώρα λοιπόν να ξεκινήσει αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει και εμείς να δώσουμε την δική μας γνωμοδότηση. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή μας για να κάνει την εισαγωγή της και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας ε, κάνω μία περιγραφή των τελευταίων μηνών. Μας Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να είναι πιο ενωμένη στο μέλλον. Ε, το περασμένο Μάρτιο πριν από το ε, κρούσμα ε, σε 40 χρόνια είχε μόλις 2.300 νεκρούς. Ε, ενώ ξέρουμε τα στοιχεία ε, για το 2014, οι γιατροί χωρίς σύνορα είπαν ότι ήταν πρωτοφανή η περίπτωση πάνω από 22.000 ε, κρούσματα και πάνω από 8.800 νεκροί. 8 χώρες πλήττονται σε τρεις υπήρους. Βέβαια κυρίως σε αυτόν τον καιρό είναι η Δυτική Αφρική η περιφέρεια που πλήττεται περισσότερο. Η επιδημία αυτή είναι και αστική, όχι μόνο στην Ήπεθρο όπως το παρελθόν και διασυνοριακή και ήταν έκτακτη ανάγκη ταυτόχρονα σε τρεις χώρες Δυτικής Αφρικής. Όπως γνωρίζετε ε, υπήρξαν και εκτός Αφρικής κάποια κρούσματα και είναι και το πρώτο στέλεχος και η πρώτη έκρηξη που ε, είδε ε, απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικό ψήφισμα. Το θέμα είναι αν εκρούσαμε το κόδωνα κινδύνου. Ε, το έκαναν οι γιατροί χωρίς σύνορα τον Απρίλιο μάλιστα του 2014. Ήταν πρωτοφανής η κρίση γιατί ήταν τα κρούσματα ταυτόχρονα σε διάφορους τόπους, σε διάφορες χώρες και πολύ γρήγορα έφτασε σε μεγάλες πόλεις. Και επίσης το στέλεχο του, ιού ήταν το πιο θανατηφόρο και το πιο επιθετικό η επιδημία ήταν τελείως εκτός ελέγχου και ουσιαστικά μία μόνο οργάνωση για τρεις χώρες σύνορα ήταν παρούσα επιτόπου και θεράπευε τους η αδυναγωγή εν πάση περιπτώσει τους ασθενείς. Χρειάστηκε μαζική παρέμφαση της Παγκόσμιας οργάνωση Υγείας και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε κυρίως έστειλαν χρήματα και πόρους, όχι μόνο λεφτά, αλλά κυρίως ε, γιατρούς, υγειονομικό, προσωπικό, ε, ανθρώπινους πόρους και ε, νοσοκομεία εκστρατείας. Άργησε όμως να περάσουμε από τις υποσχέσεις στα λόγια και προχώρησε το καλοκαίρι ε, με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τον Αύγουστο να ε, κηρύσει εθνική και παγκόσμια μάλλον επιδημία. Ε, χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια να λάβει ρόλο συντονιστικό. Το, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο δήλωσε ότι πρόκειται για απειλή. Και δυστυχώς και είναι θλιβερό αυτό και με οδύνει το λέω. Ε, για να ανάψουν εδώ πέρα τα λαμπάκια χρειάστηκε να έρθουν ε, κρούσματα στην Ευρώπη. Αλλά μέχρι τότε χάθηκαν πάρα πολλές ζωές. Η διεθνής βοήθεια έφτασε αργά και όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε για να αντιμετωπιστεί η επιδημία. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, την οποία όμως τιμώ γενικά, ε, άργησε πάρα πολύ υπερβολικά και να αντιδράσει και να ηγηθεί στην απόκριση. Θεωρώ ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα πρέπει να συντονίζει ε, και να ενοποιήσει τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για μελλοντικές εκρήξεις και κρούσματα αυτής της ασθένειας ή άλλων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να συμμετέχει. Η διεθνής ε, βοήθεια ήταν κυρίως οικονομική και πολύ λίγες ήταν οι ανθρώπινες ενισχύσεις ε, κυρίως ε, μέσω ΜΚΟ με γιατρούς και θελοντές τους. Ο έμπολα μπορεί φυσικά να εκριζωθεί, αλλά χρειάζεται να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Η επιδημία συνεχίζει ε, και χρειάζεται σωστή απάντηση. Το σημαντικότερο στόχος και η πρόκληση είναι ε, να προσαρμόζεται και η βοήθεια στην αρρώστια που αλλάζει συνεχώς. Θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και πολλοί που τηλεφωνούν για κρούσματα ενδεχόμενα, τους απαντάνε καλά να τον κρατήσετε σε απομόνωση στο σπίτι. Μα υπάρχουν ολόκληρες περιοχές όπου αρνείται κάποιος ας πούμε να αγγίξει γυναίκα τη στιγμή του τοκετού, μην τυχόν και κολλήσει έμπολα. Είναι αυτά τα πράγματα ε, ναι, λογικά σήμερα στην Ευρώπη και στην ε, Αφρική. Μας λένε ότι θα γίνουν δοκιμές για εμβόλια και πάλι κατόπιν εορτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκρισε στα τέλη του έτους περισσότερα χρήματα και περισσότερη ε, έρευνα για το έμπολα. Σωστό είναι αυτό ε, και στη Δυτική Αφρική κυρίως. Αλλά θα πρέπει όλοι να διδαχθούμε από την κρίση και από τα όσα συνέβησαν. Και βλέπω κάποια αυταρέσκεια ότι δώσαμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο λέει ε, των Ευρωπαίων καταναλωτών σε αυτή την κρίση για να καταπολεμήσουμε την έκρηξη. Θα πρέπει ο συντονισμός μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών να είναι διαφορετικό. Δεν ήταν ιδέουσα και θα πρέπει να είναι πιο ταχεία και πιο αποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα πολιτική και οικονομική εστίαση στην Αφρική και όχι μόνο για το έμπολα, πολύ περισσότερο. Θα πρέπει, όπως είπα, να είμαστε πιο ε, ευέλικτοι στην απάντηση. Τα τελευταία νέα που έμαθα σήμερα επιβεβαιώνουν ότι υποχωρεί όντως η επιδημία, αλλά δεν είναι η στιγμή τώρα να χαλαρώσουμε, γιατί υπάρχουν νέα κρούσματα, ιδιαίτερα στη Γουινέα και τη Σιέρα Λεώνα, αλλά και τη Λιβυρία. Δεν ε, ελέγχεται η επιδημία και υπάρχει δυνατότητα μετάλλαξης του ιού, όπως το Ινστιτούτο Παστέρ μόλις μας προειδοποίησε. Τα συστήματα υγείας της Γουινέας, Λιβερία και κυρίως Σιέρα Λεώνα είναι ανύπαρκτα, διαλυμένα, και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, προειδοποίησε ότι τα λεφτά τελειώνουν το Φλεβάρι, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Και ε, τέλος πιστεύω ότι η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάπως η αντανάκλαση της εύθραυστης ε, δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια κράτη-μέλη βεβαίω ήταν πιο αποτελεσματικά και κάποια άλλα πλήρης αδράνεια. αλλά ως σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στάθη στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεγητά. Και τώρα ο Σκιώδης, η Σκιώδης. Πρώτα για το ΕΛΚ κυρία Κολέν Λάγκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να καλωσορίσω την έκθεση του εισηγητού και την ανάλυση της, συμφωνώ, ε, και σε αυτά που λέει για τα διδάγματα και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν. Βεβαίω θέλω να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίω προς το παρόν μπορούμε να χαρούμε διότι ε, μειώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων. Εδώ και 42 μέρες και παραπάνω δεν υπάρχει κρούσμα πια στο Μάλι που φαίνεται ότι είναι χώρα ελεύθερη έμπολα και από τις 23 ε, πρώτου και στις Χισιαρανεώνε κάπως έχουν χαλαρώσει οι ε, περιορισμοί, αλλά δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε, να τα αναλύσουμε πάρα πολύ λεπτομερώς, να δούμε τι λάθη κάναμε, πού ήταν οι ελλείψεις και πώς μπορούμε τώρα στο μέλλον να ασχοληθούμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοια επιδημία ή κάποια αντίστοιχη. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο ιός και πώς θα πρέπει να αποτραπούν αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα που είδαμε ε, τους πρώτους μήνες. Καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω με τον εισηγητή ε, για να εξάρω όλους ε, που ρίσκαν τη ζωή τους, ψοκινδύνευσαν γιατροί, ε, νοσοκόμες, θελοντές, αρχές υγειονομικές και θα πρέπει να το πούμε κι εμείς, θα πρέπει να βρούμε νέα προϊόντα, νέα φάρμακα, νέα εμβόλια. Στον κόσμο δεν επιτρέπεται να ξαναέχουμε τέτοιες επιδημίες με τέτοια ε, απελπιστική αντίδραση. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δίνουμε καλύτερες απαντήσεις με καλύτερο συντονισμό σε τέτοιες περιπτώσεις. Συντονιστή έμπολα ορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το καλωσορίζω αυτό ρίτα, αλλά κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει και σε εθνικό επίπεδο, επιγόντως, για να δημιουργηθεί δίκτυο επικοινωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατών Μελών για το θέμα αυτό και συντονισμένη δράση. Και επίσης από τη σκοπιά της δικής μας Επιτροπής θα πρέπει να τονιστούν θέματα υγειονομικά, απόβλητα, απολύμανση, πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ε, σωστά συστήματα υπονόμων και αποχέτευσης έχουν τεράστια σημασία όλα αυτά και έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια και των Ευρωπαίων πολιτών και την υγεία τους. Θα πρέπει να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τρόπο πιο εντατικό. Και ένα τελευταίο, χωρίς αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, ε, χρειάζεται επιγόντως ε, Ευρωπαίοι Εκεί ε, ε, δεν υπάρχουν όμως ελάχιστες προδιαγραφές και ε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί να εργαστεί πλήττεται από την ασθένεια. Θα πρέπει να υπάρξει μια μέθοδος ε, εξέταση των όσων επιστρέφουν από αυτές τις περιοχές ε, για το αν έχουν προσβληθεί από έβολα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ε, σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Gracias, señor presidente. Bueno, como no puede ser de otra manera, yo también quiero comenzar agradeciendo. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του, ιδιαίτερα σε ένα θέμα που έχει αλλάξει τόσο πολύ σε τόσο λίγο καιρό και χρειάζεται ε, συνεχής ενημέρωσης και επικαιροποίηση, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα από το Δεκέμβριο και μετά. Ε, τα στοιχεία που λέει η έκθεση σήμερα ε, έχουν ξεπεραστεί και θα πρέπει να μπουν ε, τα νέα στοιχεία, τα πιο ε, ενημερωμένα. Έχω γενικές παρατηρήσεις και μία ειδική. Βεβαίως έχουμε ε, κάνει λάση και σφάλματα, το λέει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Ήταν κάπως συγκεχημένη ή μη συντονισμένη η αντίδρασή μας. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνέργεια, θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, αλλά να έχουμε και μια ε, θεώρηση όχι τόσο αρνητική, να βλέπουμε με αισιοδοξία τώρα το μέλλον για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, στην αρχή υποτίμησε ε, τα κρούσματα το Μάρτιο του 2014 και μέχρι τον Αύγουστο ήταν σε μια αδράνεια μέχρι να πει ότι είναι διεθνής η επιδημία και χρειάζεται επίγουσα ε, αντιμετώπιση. Ε, έξι μήνες χρειάστηκε για να ε, αντιδράσει. Σήμερα που σχεδόν έχει περάσει άλλο ένα εξάμεινο, πέντε μήνες, σε μπορούμε να πούμε ότι ελέγχεται σε γενικές γραμμές η επιδημία. Από τον Αύγουστο και μετά θεωρούμε ότι ήταν ε, αποτελεσματική, ικανοποιητική. Μιλάμε για τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις και τα θεσμικά όργανα. Στις 18 Ενάτου, μετά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, αλλά θα πρέπει να πω ότι άργησαν, άργησαν. Ναι. Ε, ε, οι ε, αντιδράσεις. Βέβαια, ε, στείλαμε πολλά χρήματα, 1,1 δις και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα 500 εκατομμύρια. Ε, αυτές οι οργανώσεις και οργανισμοί όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το συντονισμό διαφόρων κρατών που έχουν και διαφορετικά συμφέροντα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τόσο σημαντικά προβλήματα σε περιοχές που έχουν τόσες ανάγκες. Είμαστε επικριτικοί μεν αλλά επικοδομητικοί. Και η ίδια Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αναγνωρίσει στις 26 πρώτου ε, τα λάθη της. Τρεις έκτακτες συνεδριάσεις έχει κάνει μόνο από την ίδρυση, από τη σύστασή της. Και ε, μάλιστα ε, πάντα επρόκειτο για επιδημία. Αναγνώρισε ότι ήταν δύσκολες και πολύ διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με τα όσα είχαμε συζητήσει, συνηθίσει συγγνώμη, σε τέτοιες επιδημίες. Πρώτη φορά ξέσπασε τέτοια κρίση διεθνής ε, το είδαμε και με την γρήπη α αυτό, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω λοιπόν ότι ε, οι συστάσει, της Παγκόσμια οργάνωση Υγεία τη 26 Ιανουαρίου θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρούσα έκθεση. Και μάλιστα λέγουν τα εξή τρία. Πρώτον, σε πρώτη φάση να ενισχυθεί το σύστημα κατεπίγουσα ανάγκης του ΠΟΗ και να μεταφερθεί στην Ευρώπη και είναι σημαντικό να αναλύσουμε και να ενισχύσουμε ε, τον οργανισμό που ασχολείται με αυτά τα θέματα που παρακολουθεί και θέματα έμπολα. Έχουμε και ε, συντονιστή του έμπολα που είναι ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της πρόσβασης των νέων φαρμάκων του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι πιο ευάλωτοι λαοί και πιο ε, μειονεκτούντες. Και επίσης 800 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για να εκριζωθεί η επιδημία. Βγάλαμε πολλά διδάγματα από αυτή τη διεθνή επιδημία. Εγώ θέλω να τονίσω τα εξή δύο. Ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού και μάλιστα διεθνούς. Είναι αποτελεσματική σε αυτή την περίπτωση. Και ένα δεύτερο, τα υγειονομικά συστήματα δεν είναι πολυτέλεια. Γιατί αν υπήρξε κάτι που κατάφερε να ελέγξει περισσότερο την κρίση, ήταν ακριβώς η ισχύση όχι του υγειονομικού συστήματος κάθε χώρα. Χρειάζεται λοιπόν να εργαστούμε για να στήσουμε συστήματα υγείας σε χώρες που υπολείπονται ή που δεν είναι αρκετά ισχυρά. Πού βρισκόμαστε τώρα. Τούτων όρων λέχθεντων θα πρέπει να έχουμε ένα οδικό χάρτη για την εκρίζωση του έμπολα. Σήμερα οι επιδημιολόγοι θεωρούν ότι έχουμε περάσει σε δεύτερη φάση, ελέγχουμε τη μόλυνση και τη μετάδοση. Βεβαίως πρόκειται για ένα ιό που μεταδίδεται εύκολα, που μεταλλάσσεται εύκολα και ε, είναι δύσκολη η διάγνωση για όσους δεν γνωρίζουν ε, τα συμπτώματα του ιού ακριβώς. Γι' αυτό Το λέει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει, να ε, δεσμευτεί και εκτός από αυτό το ταμείο θα πρέπει το 20% της αναπτυξιακής βοήθειας να πηγαίνει σε βασικές υποδομές και υπηρεσίες ε, ε, κοινωνικές και δημόσιας υγείας για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Αυτό το θέμα, το υγειονομικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε αναχώρα να γίνουν αναλύσεις, μελέτες για να δούμε συγκεκριμένα πού χρειάζονται βοήθεια για να στηθούν τα συστήματα υγείας με την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και το τρίτο είναι το εμβόλιο. Έχουμε ελπιδοφόρα στοιχεία, δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο, αλλά όσο ούπο. Με ε, δημόσια κονδύλια έχει χρηματοδοτηθεί, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ρήτρα κοινωνικής ευθύνης να ε, είμαστε βέβαιοι ότι οι πιο ευάλωτοι θα έχουν πρόσβατη στο εμβόλιο, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, στη Δυτική Αφρική, γιατί είναι καινοτόμο και το εμβόλιο και ε, η θεραπεία. Είμαστε στο παραπέντε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά σημασία δεν έχει τόσο πολύ να βγει το εμβόλιο, αλλά να ε, έχουν πρόσβαση άνθρωποι για να εκριζωθεί η νόσος. Με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα, για να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο για όλους τους ασθενείς. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πιέσουμε τη διεθνή κοινότητα και τα θεσμικά όργανα για να κάνουμε πραγματικότητα την εκρίζωση αυτής της νόσου που φαίνεται ότι είναι κάτι το εφικτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πιέτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον εισηγητή μας για την ποιότητα της προσπάθειας την οποία έχει κάνει. Βέβαια από τότε έχουν ε, συμβεί αρκετά πράγματα, θα πρέπει κάπως να ενημερώσουμε ε, την ε, πρόταση. Αυτό συνδέεται κυρίως με την έρευνα ε, η οποία έχει προχωρήσει σε σχέση με τον ιό εμπόλα. Έχουμε περάσει σε ένα εμβόλιο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προωθηθεί αρκετά και βρισκόμαστε στις κλινικές δοκιμές που είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την πλήρη χρήση αυτών των εμβολίων θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας και των Ηνωμένων Εθνών για να εκριζώσουμε τον ιό αυτό όπως το κάναμε και για άλλες ασθένειες στο παρελθόν. Χρειάζονται όμως ε, ε, μαζικοί εμβολιασμοί και αυτό δημιουργεί οικονομικά ε, ερωτηματικά. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε στο μέλλον να βοηθήσουμε οικονομικά τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Σύνεπως, η εκρίζωση του ιού αυτού δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο μέσω ε, μέτρων ε, πρόληψης. Πρόληψης ε, ενεργής, δραστήριας, ιδιαίτερα για τους πλέον εκτεθειμένους πληθυσμούς. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά Ελπίζω οι παρατηρήσεις αυτές για τη βοήθεια η οποία θα πρέπει να δοθεί στις συγκεκριμένες χώρες για τον έλεγχο της επιδημίας εμπόλα να γίνει πραγματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να ξεχάσουν ότι πρόκειται για φτωχές χώρες, χώρες ε, οι οποίες ε, πολλές από αυτές βρίσκονται σε σύγκρουση με γειτονικές χώρες ή εσωτερικού τύπου εμφύλιες σειράξεις και θα πρέπει να συνεχίσουμε την οικονομική βοήθεια προς αυτές. Μπέρντερ για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, ε, τον εισηγητή συγγνώμη, για την προσπάθειά του. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στην τύχη των θυμάτων και στη τύχη των οικογενειών τους. Υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα τα οποία μπορούμε να καταλήξουμε εδώ στην Ευρώπη. Ε, είναι σαφές ότι αντιδράσαμε με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η απειλή για την Ευρώπη παραμένει σημαντική, αλλά παρόλα αυτά δεν αντιδράσαμε έγκαιρα. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε στο μέλλον με υψηλότερη ταχύτητα. Έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ οι χώρες αυτές της Δυτικής Αφρικής και για λόγους πολιτισμικούς οι χώρες αυτές έπρεπε να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ε, το θέμα των θανάτων και γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η εποχή αυτή και είναι για τις οικογένειες που υποφέρουν από τις απώλειες των δικών τους. Έχουν υπάρξει κάποια βήματα πάντως. Ε, ένα τμήμα της νέας τεχνολογίας ε, της έχει βοηθήσει ε, συνεχή μηνύματα στο τηλέφωνο σαν παράδειγμα για να πλένουν τα χέρια τους κτλ. Είναι ένας τρόπος που δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε κοντά στους ανθρώπους αυτούς πριν 10 χρόνια. Οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, ποιος να το πίστευε. Είναι όμως καρπός ε, πράγματι συνεργασίας και το Ινστιτούτο στο οποίο δούλευα και στην Οξφόρδη εξακολουθεί να ασχολείται με την φυματίωση και με την ελονοσία και κάποια από τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε εκεί ε, μεταφέρθηκαν στην έρευνα για τον εμπόλα. Αυτή η έρευνα λοιπόν γίνεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πάρα πολύ συχνά λοιπόν οι μεγάλες χώρες ε, ε, δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρα σε αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες αλλά μπορούν να τις πάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ωφέλεια για αυτές. Η δύσκολη πλευρά πλέον τώρα αυτής της ασθένειας είναι ότι τα πρώτα θύματα ήταν οι νοσηλευτές. Στη Λιβερία ιδιαίτερα όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή υπήρχαν μόνο 51 γιατροί και στη Σιέρα Λεόνε με 6 εκατομμύρια πληθυσμό ήταν 106 γιατροί. Συνεπώς λοιπόν ε, οι γιατροί και οι νοσοκόμες ήταν στην πρώτη γραμμή και ε, υπήρξαν πάρα πολλές απώλειες. Γιατί υπήρχαν τόσοι λίγοι γιατροί. Ε, γιατί πράγματι εμείς τους παίρνουμε στη Δύση, παίρνουμε τα, τους καλύτερους γιατρούς από την περιοχή αυτή στη Δύση. Ενώ πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε να μπορούν να δουλεύουν στις χώρες τους και να μην έρχονται όλοι στην Ευρώπη ή στην Αμερική αναζητώντας βέβαια τους υψηλότερους ε, μισθούς, κάτι το οποίο είναι δίκοπο μαχαίρι για τις χώρες προέλευσης. Ένας άλλος τομέας στον οποίο ε, κάναμε λάθος είναι ε, τα μεγάλα νοσοκομεία αντίθετα με τις μικρές κλινικές. Τα μεγάλα νοσοκομεία δεν μπόρεσαν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις. Και αυτό γιατί η νέα τεχνολογία που είναι διαθέσιμη είναι πραγματικά πολλά υποσχόμενη. Ε, και μέσω των τηλεφωνικών δικτύων είδα παραδείγματα στήριξης των μικρών νοσοκομείων ε, που παραγγέλουν τα φάρμακα και τον εξοπλισμό τους με μεγάλη ταχύτητα και ε, χωρίς κινδύνους. Και τέλος το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και ποια είναι τα συμπεράσματα, η κληρονομιά αυτής της κατάστασης. Οι χώρες αυτές είναι σε δύσκολη κατάσταση πια. Έχασαν καλλιέργειες, σοβιές γιατί δεν φύτεψαν. Έχασαν πάρα πολλούς γιατρούς, έχασαν πάρα πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μικρά μαγαζάκια, οι μικροί μεταφορείς έχουν χάσει ε, πρόσωπα μέσα κτλ. Αυτό θα απαιτήσει πάρα πολλά χρόνια. Άλλα οικονομικά προγράμματα όπως οι μαγουλάδες ή η πολυμελίτιδα έχουν διακοπεί και υπάρχει μια ανάκαμψη των ασθενειών αυτών που νομίζαμε ότι είχαμε στο παρελθόν ελέγξει. Και φυσικά έχουμε και την βαριά κληρονομιά των ορφανών που επιβίωσαν σε κατεστραμμένες κοινότητες και απαιτείται μακροπρόθεσμη βοήθεια προς τις χώρες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε και τον αστικό χαρακτήρα αυτών των προβλημάτων. Η Τενεκεδουπόλης είναι πραγματικά χώρος εκόλαψης ιδανικός για τις ασθένειες αυτές και αυτό φάνηκε από όλες τις ιατρικές παρεμβάσεις. Τελειώνοντας θα πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι αιτίες του προβλήματος αυτού. Θεωρείται ότι η ασθένεια αυτή ήρθε από την κατανάλωση άγριων ζώων. Είναι μια πηγή πρωτεΐνης ε, από την οποία εξαρτώνται οι αφρικανικές χώρες. Ε, δεν είναι αηφόρος βέβαια και επίσης στέλνονται και στην Ευρώπη σε τεράστιες ποσότητες. Σήμερα ακούσαμε από έναν από τους ομιλητές μας ότι η Ευρώπη είναι τόσο ισχυρή όσο το ασθενέστερό της σημείο και η εισαγωγή παρανόμως κρέατος αγρίων ζώων είναι τρομερός κίνδυνος και θα πρέπει λοιπόν εδώ να προσέξουμε. Θα καταθέσω τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος νομίζω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε και την οποία εκτιμούμε δεόντως. Θα συμφωνήσω μαζί του όταν λέει ότι πέρα από τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται στην Αφρική για την απομόνωση του ιού, οι τελευταίες εξημίσεις ε, του διεθνούς, της Διεθνούς Οργάνωσης ε, ε, Υγείας ε, έδειξαν ότι και σε μεγάλες χώρες υπήρξαν πολλά προβλήματα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών, ιδιαίτερα σε επίπεδο νοσοκομιακών δομών. Δεν πετύχαμε τον στόχο, ε, σαν παράδειγμα, ε, της προμήθειας εξοπλισμού προστασίας για τις 14 χώρες που έχουν εκτεθεί στη συγκεκριμένη μορφή του ιού. Πάρα πολλέ ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια. Να σα υπενθυμίσω και την οργάνωση Emergency, η οποία, στην οποία δεν αναφέρθηκε κανείς, ήταν στην πρώτη γραμμή στα πλαίσια της καταπολέμησης του εμπόλα. Να προσθέσω ένα σημείο μόνο το οποίο ε, κατ' εμέ θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Την ανάγκη να απομονώσουμε τον ιό αυτό αλλά να μην απομονώσουμε τους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να του δώσουμε εγγυήσεις ασφάλειας, ε, να το βοηθήσουμε φυσικά σε επίπεδο υγείας, παροχής υπηρεσιών υγείας, μεταφοράς άμεσα εφόσον διαπιστωθεί έκθεση στην ασθένεια κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που το ζήτησαν. Η κυρία σραιερ Ευχαριστώ. Τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, ε, έκανα την πρώτη ερώτηση και γι' αυτό ξανά να κάνω και τις επόμενες. Ευχαριστώ τους συγητές. Το τελευταίο ε, διήμερο για τρίτη φορά συζητούμε και στην ΑΚΕ και στην ΕΜΒΕ. Είναι σημαντικό το θέμα. Ε, το θέμα είναι να δούμε τι διδάγματα θα βγάλουμε και πώς η Ευρώπη αντέδρασε. Εκ των υστέρων φυσικά όλοι τα ξέρουμε καλύτερα. Βεβαίως θα πρέπει να βγάλουμε μαθήματα όχι μόνο από την έμπολα αλλά και από την φυματίωση, το είπατε και εσείς πρόεδρε και έπονται άλλες ασθένειες πολύ σοβαρότερες. Είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε αρκετά χρήματα στην άκρη και στην Επιτροπή μας μέσω οργανισμών ή δεν ξέρω ε, για αυτούς τους σκοπούς. Περί αυτών πρόκειται. Εκεί πονάει ακριβώς ε, το θέμα. Έχουμε τόσα ψηφίσματα υπογράψει και το Σεπτέμβριο στο Στρασβουρού και συμμετείχα κι εγώ και είπαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί επαρχή σηματοδότηση και βρήκαμε 500 εκατομμύρια, αλλά ήταν περισσότερες οι ανάγκες. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και τέλος δύο σύντομες ερωτήσεις. Είχα ρωτήσει και τον Επίτροπο. Υπάρχουν πάρα πολλά ορφανά και χρειάζονται χρήματα για να χτιστούν ορφανοτροφία. Συγκεκριμένα μπορεί κάποιο να μου πει ότι έγινε αυτό. Ένα. Και δεύτερον, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όχι μόνο τους εθελοντές και τα κράτη-μέλη. Και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που έγιναν πάρα πολλά πράγματα και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε. Μιλάμε για το καθαρό νερό και να πλένουν τα χέρια τους. Για πηγαίνετε στις χώρες εκεί να βρείτε καθαρό νερό. Και όταν έχεις καθαρό νερό το πίνεις μάλλον και δεν πλένεις τα χέρια σου με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία μου. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο. Γι' αυτό θα τον δώσω στον Μάρκ Σπρίγκερ, εκτελεστικό διευθυντή του ΩΣΑ, ECDC. E In fact, the, the report of the, the rapporteur... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι λίγο θλιβερή η έκθεση του εισηγητή, αλλά είναι αληθινή και συμφωνώ και με τους υπόλοιπους. Δεν είναι πολύ θετικά όλα αυτά. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να πάρουμε μαθήματα από αυτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός μας έχει πέντε ομάδες που δουλεύουν στη Γουινέα με επιδημιολόγους και προσπαθούν να δημιουργήσουν τοπικά συστήματα οργάνωσης αντιμετώπισης της ασθενείας και δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα όπως έλλειψη καυσίμων ας πούμε και δεν μπορούμε έτσι να φτάσουμε σε μακρινές περιοχές. Ε, επίσης μπορεί να υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Δεν είναι πάντα εύκολο για τις ομάδες μας να φτάσουν στις απομακρυσμένες περιοχές. Πολύ δύσκολο λοιπόν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θετικό είναι όμως ότι η Αφρικανική Ένωση θα ήθελε ή μάλλον αποφάσισε να ορίσει ένα Αφρικανικό κέντρο για έλεγχο επιδημιών και ήρθαμε σε επαφή όχι μόνο με το Σύντηση στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και μας διότι ίσως οι ευρωπαϊκές δομές να μοιάζουν περισσότερο με τις αφρικανικές όπου Υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα κράτη. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με την Αφρικανική Ένωση μέσω της εκπροσώπησης της Ένωσης και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους υποστηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε για να καθορίσουν ένα πιο βιώσιμο τρόπο ελέγχου των κολλητικών ασθενειών. Λιμόδι. Λιμόδι. Είναι πολύ εύκολο να ψέξουμε τον ΠΟΗ, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μην βιάζεστε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέγομαι Δόκτωρ Φίλιπ Μόλλερ και εργάζομαι στην ΕΚΟ. Ως γιατρός εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι πρέπει να γίνονται νεκροψίες αλλά επίσης πρέπει να περιμένουμε να πεθάνει πρώτα ο ασθενής. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να πάρουμε στρατηγικά μαθήματα ή μαθήματα στρατηγικής. Εν τω μεταξύ κάναμε πολλά λάθη μέχρι να μάθουμε να πάρουμε τα μαθήματα τακτικής που χρειαζόμαστε. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, η επιδημία συνεχίζεται και πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας πρώτον στη σταμάτημά της. Μέχρι ενός σημείου βέβαια δεν πρέπει να υπερβάλλουμε στην αυτοκριτική μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν γενικότερα έχουν πετύχει και μερικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη. Στην ΕΚΟ χρηματοδοτούσαμε τον ΠΟΗ, τον Ερυθρό Σταυρό κλπ. Τα αρχίσαμε να τα χρηματοδοτούμε όλα αυτά μέσα σε μια εβδομάδα. Οι συνάδελφοι από την ΤΕΦΚΟ κινητοποιήθηκαν επιτόπου στη Γουινέα μέσα σε μια εβδομάδα Στείλαμε εμπειρογνώμονες επίσης μέσα σε μια εβδομάδα. Επίσης προσπαθήσαμε στη χρηματοδότησή μας να στηρίξουμε και τα κέντρα αντιμετώπισης ασθενειών και άλλων εκτός εμπόλα. Το κέντρο άμεσης αντιμετώπισης της Ένωσης οργάνωσε πολλές συναντήσεις και συνεδριάσεις από τις πρώτες εβδομάδες στις υπηρεσίες της Κομισιόν και μετά και στις χώρες μέλη και μπορώ να σας πω ότι καθημερινά γίνονταν τέτοιες συναντήσεις και πολλές χώρες μέλη έχουν συμμετάσχει ανελιπώς από την αρχή της επιδημίας και ακόμη συνεχίζουν. Τις συνεδριάσεις αυτές τις έχουμε ανοιχτέ και στον ΟΗΕ. Και έρχονται και αυτοί μία φορά τη βδομάδα. Επίσης έχουμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης που επιτρέπει από υπηρεσίες του ΟΗΕ να ζητούν ότι μπορούμε να περάσουμε στη συνέχεια στα κράτη-μέλη. Επίσης, συστήσαμε, έκαναμε μεγάλη, με μεγάλη προσπάθεια το σύστημα Medivac που επιτρέπει σε εκπατρισμένους προσωπικό διεθνών οργανισμών και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη σε περίπτωση προσβολής μόλυνσης. Όλα αυτά έχουν αποφέρει αποτελέσματα και τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι μαζί με τους συναδέλφους μας με τις άλλες γενικές διευθύνσεις ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου οργανώσαμε μια διεθνή διάσκεψη για την επιδημία του έμπολα ε, ήρθαν, προσήλθαν οι περισσότερες χώρες το ίδιο έγινε και στις 12 Δεκεμβρίου και μάλλον θα ξέρετε ότι και στις 3 Μαρτίου θα γίνει μια τρίτη τέτοια διεθνής υψηλού επίπεδου διάσκεψη για την επιδημία του έμπολα για να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει για να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να ανακάμψουν. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια ήμασταν λιγότερο επιτυχείς και ο κύριος τομέας όπου ως συντονιστής των προσπαθειών θεώρησα ότι είχαμε λήψεις είναι το ότι αποτυχίες είναι το ότι δεν δημιουργήσαμε ένα μόνιμο σώμα ιατρικού προσωπικού που να μπορεί να σταλεί όπου χρειαζόταν. Οι συνάδελφοι του ECD είναι μόνο 350. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, το κέντρο ελέγχου των επιδημών δρυμιών στι ΗΠΑ Πολιτείες έχει 5.000. 15.000. Και τελικά χρειάστηκε ένα προσωρινό υποτυπώδες σύστημα να οργανωθεί και αυτό ίσως είναι ένα μάθημα που μπορούμε να πάρουμε. Η Γαλλία και η Γερμανία συνέγραψαν μία λευκή βίβλο για να δουν αν μπορεί να οργανωθεί κάτι τέτοιο κάποιο απόθεμα κατά κάποιον τρόπο ιατρικού προσωπικού. Πολλά μαθήματα λοιπόν μπορούμε να πάρουμε και είναι πολύ χρήσιμο αυτό που εξετάζει σήμερα το Κοινοβούλιο, αλλά το κύριο είναι να καταπολεμηθεί η επιδημία. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο συνάδελφός μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι την Τιέβερσε. Είμαι τμήματάρχη για τη Δυτική Αφρική. Όπως ακούσατε, η μεγάλη συνάντηση θα οργανωθεί για την 3η Μαρτίου, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν την κατάσταση στις τρεις χώρες που έχουν φυγεί κυρίως από τον Εμπόλα. Είναι τρεις χώρες έφραστες μετά από κρίσεις, μετά από συγκρούσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα λοιπόν στις χώρες αυτές. Υπάρχει έλλειψη διακυβέρνησης, υπάρχει κακή διακυβέρνηση και γενικά έχουν και προβλήματα πολύ σοβαρά χρηματοδότησης ε, οι χώρες αυτές. Λοιπόν, τα χρήματα είναι μερικές φορές η αρχή της απάντησης στην περίοδο μετά την κρίση που θα πρέπει να προχωρήσουμε μαζί με τις κυβερνήσεις τους. Συνδέεται με τα προγράμματα των τριών κυβερνήσεων. Είναι σαφές ότι και η Παγκόσμια Τράπεζα και εμείς και τα Ηνωμένα Έθνη θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη Γουινέα, τη Σχέρα και τη Λιβερία μέσω πρόθεσμα προβλέπεται η κοινωνική τομής, η βασική, ε, να, να υποστηριχθούν στη Σιέρα Λεόνε και στη Λιβερία η εκπαίδευση και στην Γουινέα η υγεία. Η ασφάλεια βέβαια, η υγεία και η ε, αντοχή είναι βασικό θέμα. Κάποιες λοιπόν αναλύσεις τις οποίες έχουμε κάνει σε σχέση με τον εύπαστο χαρακτήρα των χωρών αυτών είναι συμβατές με τις παρεμβάσεις μας μετά από την κρίση του εμπόλα. Μία δράση την οποία έχει ξεκινήσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ενισχύσει δημοσιονομικά τη Σιέρα Λεόνε και την εμπόλα γιατί η κρίση αυτή δημιούργησε τεράστια ελλείμματα που θέτουν σε, λειτουργή, αμφισβήτηση την λειτουργία του κράτους και θα ήταν καταστροφικό να βρεθούμε σε ένα σενάριο όπως την κεντροαφρικανική δημοκρατία με εξαφάνιση των κρατικών δομών. Βοηθήσαμε λοιπόν τη Λιβερία και του Σιέρα να διατηρήσουν τις κρατικές δομές μέσα από άμεσες δημοσιονομικές ενισχύσεις με σημαντικά ποσά τα οποία δόθηκαν το 2014 μετά από την κρίση του εμπόλα. 30 εκατομμύρια στην Λιβερία και 22,6 στη Σιέρα Λεόνε. Τέλος, έχουμε τακτικές αποστολές οι οποίες εργάζονται εκεί και στον τομέα της υγείας και στις χώρες όπου δεν υπάρχουν οργανωμένες δομές υποδοχής των συστημάτων υγείας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κρίση του εμπόλα που χρηματοδοτούνται και από επιμέρους ε, κράτη-μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο στη Σιέρα Λεόνε και οι Ηνωμένε Πολιτείε στη Λιβερία. Υπάρχει μια αποστολή την οποία είχαμε στείλει και επεστρέφει σήμερα από την Γουινέα Κονακρή για, τους, για τα ορφανά παιδιά. Υπάρχουν ήδη κάποια χρήματα διαθέσιμα σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνδέσουμε το κατεπήγον με την ανάπτυξη. Και έτσι νομίζω ότι ε, θα ανταποκριθούμε στα αιτήματα της χώρας και των ΜΚΟ. Να συμπληρώσω ότι τα πράγματα δεν είναι όλα βέβαια πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά έχουμε ενισχύσει ε, τον συντονισμό μας, έχουμε στείλει ταχύτατα υγειονομικό προσωπικό και νομίζω ότι και σε συνεργασία με τις άλλες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδυαστήκαμε για να έχουμε αυτό που ονομάζουμε στην αγγλική comprehensive approach. Με τα μέσα βέβαια τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας και με χρονοδιαγράμματα διαφορετικά ανάλογα με τα μέσα. Κάποια απαιτούν περισσότερο χρόνο αλλά έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια στη Γουινέα Κονακρή σαν παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εμπλακεί στον τομέα της υγείας, είμαστε η πρώτη δωρήτρια δύναμη μέχρι το 2020 τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ κύριε Βερσέ, θα ξαναδώσω το λόγο στον γνωμοδότη μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες και τις γνώμες όλων των συναδέλφων. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία για την συνεισφορά τους. Νομίζω ότι μπορεί να διαφέρουμε σε ορισμένες από τις μορφές της απάντησης την οποία θα πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες αυτές. Αλλά οι διαφορές αυτές είναι ελεγχόμενες. Αυτό το οποίο νομίζω είναι βασικό είναι να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχόμεθα και νομίζω ότι συμπίπτουμε πλήρως όταν συζητάμε το θέμα αυτό με επικοδομητικό πνεύμα και με πρόθυμο τρόπο. Υπάρχουν όπως είπα διαφορετικές ιδέες οι οποίες ε, έχουν σχέση με το συντονισμό, με την ενημέρωση, με την σωστή επικοινωνία, ε, με την ιδέα να, να υπάρξει μια θέση συντονιστή για τον εμπόλα, ε, για τον συγκεκριμένο ιό θα μπορούσε να γίνει αυτό ίσως στο παρελθόν και για άλλες ασθένειες και νομίζω ότι τα μαθήματα που έχουμε πάρει από άλλες λοιμώδεις ασθένειες μπορεί να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τον συγκεκριμένο ιό. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει πολύ καλός συντονισμός ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την, τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας νομίζω ότι τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι πριν λίγο, αναγνωρίζουμε την εργασία που έχει κάνει ο ΠΟΗ, όπως επίσης και όλες οι άλλες οργανώσεις και αυτό φαίνεται και στα δημοσιονομικά μας. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ε, ε, επικοδομητικοί για να μάθουμε ακριβώς και το τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Το μέλλον για τις χώρες αυτές είναι ιδιαίτερος περίπλοκο, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε πλήρως. Θα πρέπει φυσικά να προσέξουμε το τι γίνεται στις απομεμακρυσμένες περιοχές όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει κανείς εκεί και ταυτόχρονα η κατάσταση ε, που στις περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις ένοπλες είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Αλλά πάντως ε, μπορούμε να είμαστε πιο απαιτητικοί και να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε κάνει αρκετά με τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να έχουμε όμως και περισσότερα μέσα, νεότερα μέσα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσει να αξιολογήσει τις καταστάσεις στις τρεις αυτές χώρες, τη Σιέρα Λεόνε, τη Γουινέα και τη Λιβερία. Να αξιολογήσουμε λοιπόν την κατάσταση σε κάθε μία χώρα μετά από επιτόπια εξέταση. Φυσικά υπάρχει ανάγκη να περιορίσουμε τον ιό αυτό και να τον ελέγξουμε ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες είναι οι πιο απειλούμενες. Να δούμε και με τα θύματα επίσης, τις γυναίκες, τα ορφανά και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε κυρίως τα συστήματα τα τοπικά υγείας, να τα ενισχύσουμε τα μέσα τα οποία υπάρχουν και να τους δώσουμε και νέα μέσα έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους εμπλεκομένους και αυτό προς όφελος όλων. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο για την ποιότητα της παρεμβάσεώς τους τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Κατάθεση τροπολογιών 10 Φεβρουαρίου, 12 μεσημβρινή. Ε, η ψηφοφορία 26 Μαρτίου στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Ανάπτυξης 13 και 14 Ιουλίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το σημείο 20. Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τις κλινικές δοκιμές που γίνονται σε τρίτες χώρες. Πρόκειται για ένα θέμα που τέθηκε ε, στην ημερήσια διάταξη μετά από αίτημα του Πέτερ Λίζε και του δίνω αμέσως το λόγο. vielen Dank, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Περί τίνος πρόκειται. Το Δεκέμβριο δημοσιεύτηκε ότι μία εταιρεία ονόματι τη GFK Bioscience έχει κάνει κλινικές δοκιμές στην Ινδία παραβιάζοντας μαζικότατα τους κανόνες. Εδώ και χρόνια από την έκθεση της Γκλένης Βίλμοτς και μετά θυμάστε ε, είχαμε την εξή κατάσταση. κλινικές δοκιμές όταν γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έγκριση νέων φαρμάκων θα πρέπει να γίνονται βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων. Και πριν από πολλά χρόνια ακούγαμε ότι δεν γίνεται πάντα κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πριν από μία τριετία εμείς ασχοληθήκαμε και με τις κλινικές δοκιμές στις τρίτες χώρες και καλήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προσέξει πάρα πολύ. Και το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε απέναντι σε αυτές τις απάτες είναι η αφαίρεση της άδεια. Γι' αυτό την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε, όχι για όλα τα προϊόντα, ε, όπου ήταν παράνομες ε, δοκιμές, αλλά κυρίως για τα γενώσιμα σε διάφορες εταιρείες που μας εξαπάτησαν, τους αφαίρεσε την άδεια. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και θέλω να συγχαρώ τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την να ακολουθήσει αυτή τη σύσταση. Τώρα θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το ιστορικό και το υπόβαθρο. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τον ΕΟΦ. Στη γνωμοδότηση του ΕΟΦ αναφέρεται ότι αυτό δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία των ασθενών. Αυτό πόθεν. Για ποιο λόγο τότε κάνουμε κλινικές δοκιμές. Δοκιμέ γίνονται όταν πρέπει να ψάξει ένα φάρμακο ε, αν πειράζει τους ασθενεί. Εάν δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο, τότε γιατί κάνουν απάτες. Και αν δεν έχει και συνέπειες για την υγεία των ασθενών, γιατί γίνονται όλε αυτές οι δοκιμέ. Αλλά νομίζω μπορεί να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Ρης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας. Έχετε το λόγο κύριε μου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Παρουσιάσαμε δύο, θα κάνουμε δύο παρουσιάσεις. Για το γενικότερο πλαίσιο που καθορίσαμε για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, η μία και η άλλη πιο λεπτομερής για το πώς θα γίνει αυτό. Αρχίζοντας λοιπόν από τις ε, οδηγίες και τους κανονισμούς. Δημιουργήθηκαν νέοι κανονισμοί και κανόνες. Πήραμε μερικές σημαντικές αποφάσεις. Πρώτον να συγκεντρώσουμε την υποβολή των αιτήσεων σε ένα και μόνο ενωσιακό ιστό. Οι γλώσσες θα καθορίζονται από την κάθε χώρα που ενδιαφέρεται. Έχουμε ένα μηχανισμό συνεννόησης και συντονισμού Και τέλος, αυτόν τον διαβουλεύονται και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και οι καθηγητέ. Η Τράπεζα Δεδομένων και ο Ιστοσελίδα θα δημιουργηθούν από την ΕΜΑ σε συνεργασία με την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Αυτά δεν έχουν τελειώσει ακόμα, υπάρχουν ακόμη λειτουργούν ομάδες εργασίας για να τα τελειώσουν και γίνεται και δημόσια διαβούλευση που άρχισε πριν από μερικές εβδομάδες. Η εφαρμογή του εργαλείου αυτού θα αρχίσει τέλη του 16 αρχές του 17 Το σημαντικό θέμα που ανέφερε και ο Δόκτωρ Λίζε είναι να γίνουν κλινικές δοκιμές διότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνονται με βάση το πρωτόκολλο, τον ενομισμένο πρωτόκολλο που δέχονται όλοι και σύμφωνα με τις αρχές των βελτίστων κλινικών πρακτικών. Αυτά είναι πρότυπα που έχουν καθιερωθεί διεθνώ. και γίνει δεκτά. Τώρα φτάνουμε στην υποβολή των δεδομένων από τις κλινικές δοκιμές. Εκτός ένωσης, οι κλινικές δοκιμές πρέπει να συμφωνούν με κανόνες ισότιμους με εκείνους που ισχύουν στην Ένωση και πρέπει να υποβάλλονται σε ένα μητρό του ΠΟΗ και να δημοσιεύονται σε περιοδικά που τα ελέγχουν οι συνάδελφοι. Η χρησιμοποίηση δεδομένων από αυτές τις δοκιμές χρειάζεται άδεια Όπως είπα, οι δοκιμές πρέπει να γίνονται με βάση τα διεθνή πρότυπα ισότιμα με τις Ένωσης και πρέπει να γίνονται επίσης σύμφωνα και με ε, δεοντολογικές αρχές με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, όχι τους μέλλοντες, αλλά τους ισχύοντες. Τώρα, πώς θα μπορούσαμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Ο συνάδελφος μου θα σας τα πει σε λεπτομέρειες. Οι έλεγχοι στους τόπους που γίνονται οι δοκιμές και σε Ένωση και σε τρίτες χώρες θα γίνονται από τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε ενωσιακούς επόπτες. Τα κράτη-μέλη θα πληροφορούν για τη συμπλήρωση των δεδομένων και για τις, τους ελέγχους η ΕΜΑ θα συντονίζει τους ελέγχους αυτούς για να χρησιμοποιούνται οι πόροι πιο αποτελεσματικά ανάλογα με το πόσους ελπόπτες έχουμε και οι εκθέσεις τους θα φορτώνονται, θα συμπληρώνουν την τράπεζα των δεδομένων. Σε κάθε διμερή συνάντηση που έχουμε με τρίτη χώρα από τον Νοέμβριο, όπως τον Νοέμβριο με την Κίνα, θα το θέτουμε αυτό το θέμα και θα το πληροφορούμε και με την Κίνα και με άλλες. Εκεί εξηγούμε τις μεθόδους μας, αλλά επίσης θα ήθελα να σας πω ότι Όλα αυτά άρχισαν με βάση έναν γαλλικό έλεγχο τον οποίο, τον οποίο υπέβαλε η Γαλλία στην Κομισιόνα. Το νέο σύστημα θα κάνει μόνο του τους ελέγχους, δηλαδή θα παρακολουθούνται και τα συστήματα εποπτείας των χωρών μελών και σε τρίτες χώρες και οι δημοσιονομικοί έλεγχη θα συντονίζονται Θα τα ξαναπούν όλα αυτά με τα κράτη-μέλη βέβαια και οι δημοσιονομικοί όπως είπα έλεγχοι θα γνωστοποιούνται δημόσια και θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματά τους. Τέλος, η ενωσιακή έλεγχη θα γίνονται από την υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρικής και θα αφορούν και ορισμένα φαρμακολογικά συστατικά. Πρέπει να βρούμε γενικώ τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. έρθω από την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ πολύ. Ο δόκτωρ Σουίνι. Χαίρετε. Καλησπέρα σας κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και τον Δόκτωρα Λίζα για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνουμε σήμερα εδώ αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα πρώτα να σας δώσω τη γενική εικόνα. Υπάρχει μια κεντροποιημένη διαδικασία, κλινικές δοκιμές ανατίθενται, θα σας πω με ποιο τρόπο, μετά πώς γίνεται ο έλεγχος και πώς γίνεται ο έλεγχος για τα γενώσιμα φάρμακα, που είναι το θέμα της εταιρεία GVK Biosciences και πώς γίνονται οι μελέτες ε, ε, ισοδυναμίας ε, στι κλινικές δοκιμές και θα περάσω στον έλεγχο και την επιθεώρηση του GVK και πώς παραπέμφθηκε στην ε, ε, αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και θα σας αναφέρω στη συνέχεια τα μελλοντικά βήματα που προτείνουμε. Στην επόμενη διαφάνεια ε, είναι καινοτόματα προϊόντα στα οποία ε, γίνονται κλινικές δοκιμές ή αιτήσει, 10 με 100 δοκιμές ε, ε, σε γενική... Άλλο, τα γενό σημαίνει διαφορετική η κατάσταση. Είναι μία με τρεις κλινικές δοκιμές και 24 οι ασθενείς που είναι κυρίως εθελοντές οι ε, περισσότερες αιτήσει για τα γενώσιμα υποβάλλονται στα κράτη-μέλη για την εθνική αδειοδότηση, η αμοιβαία αναγνώριση ή τις αποκεντρωμένες διαδικασίες για την εναρμόνιση των αδειών μεταξύ των κρατών μελών. Και τέλος, όπως είπε και ο συνάδελφος Δοκτωρής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επιθεωρήσεις ίδιε γίνονται από επιθεωρητές των κρατών μελών και των αρμοδίων αρχών με τις οποίες συνεργαζόμαστε στενά. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε και πάλι στοιχεία για τις κλινικές δοκιμές ευρείας κλίμακας για τα καινοτόμα φάρμακα που υποβάλλονται στον οργανισμό μας. Βλέπετε ε, ότι με πράσινο εμφανίζονται οι χώρες τις οποίες ε, έχουν ε, χρησιμοποιηθεί ασθενείς, εθελοντές που δήλωσαν και 35% περίπου των ασθενών προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική, Καναδά και Ηνωμένε Πολιτείες 37% περίπου στην Ευρώπη και το υπόλοιπο στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. 9% στη Λατινική Αμερική, 2,5% στην Αφρική, 4,7% στη Ρωσία, 9,5% στη Νότιο Ανατολική Ασία. Στην Ινδία, για παράδειγμα, οι δοκιμές εκπροσωπούν μόλις 2% του συνόλου. Θα επανέλθω όμως στο ρόλο που παίζουν στις ε, μελέτες και δοκιμές βιοϊσοδυναμίας. Μπορεί να σας ε, φαίνεται λίγο το 2% αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις δοκιμές. Εδώ βλέπετε τα ίδια στοιχεία σε άλλη γραφική παράσταση. Από το 2005 μέχρι το 2013 εξελίξεις ε, παρελθούς δεκαετίας ε, η κίτρινη γραμμή είναι εκτός, η καμπύλη μας εκτός ε, Αμερικής και Ευρώπης, η κόκκινη είναι η Βόρεια Αμερική και η μπλε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Βλέπουμε ότι κατά τη δεκάτη αυτή υπάρχει αύξηση σε όλες τις περιφέρειες με κύμανση αναέτος, αλλά πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια ήταν λιγότερη η αύξηση ε, στις κλινικές δοκιμές εκτός Ευρώπης και Αμερικής. Βέβαια αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τη διακύμανση στις ε, εγκρίσει. Τι μας λέει αυτή η κατάσταση. Συνολικά την τελευταία δεκαετία έχουμε 1,2 ε, εκατομμύρια ασθενεί μέχρι το 2013 και για πέρυσι αναμένονται 200.000 κάτι τέτοιο στοιχεία ασθενών. Και οι ασθενεί αυτοί προέρχονται από 100.000 δοκιμές σε 107 χώρες. Βέβαια μερικές από τις δοκιμές αυτές μπορεί να είναι περιορισμένες. Ε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, αλλά ε, συνολικά είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. 635 νέες αιτήσει για άδεια και σε σχέση με αυτές έχουν γίνει επιθεωρήσεις για καλές κλινικές πρακτικές. 419 ε, στον αριθμό από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων γίνεται ο συντονισμός και ο έλεγχος από τους Ευρωπαίους επιθεωρητές στην Ευρώπη στην ίδια περίοδο ήταν 5.000 οι επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων των 419 για λογαριασμό του συστήματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων αλλά και για μελέτες βιοϊσοδυναμίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ε, εθνικές ή αποκεντρωμένες αιτήσει αδειοδότησης και έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά. Κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται και οι επιθεωρήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι κλινικές δοκιμές που γίνονται εδώ από τις οποίες εξαρτώμεθα και εμείς και οι υπόλοιποι στον κόσμο για τις εγκρίσεις γίνονται με τρόπο σωστό και με καλές πρακτικές και οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που έχουμε ορίσει τηρούνται. Η επόμενη διαφάνεια σας δείχνει την εξέλιξη ε, των επιθεωρήσεων και ελέγχων καλών κλινικών πρακτικών από το 2000 στα αριστερά μέχρι το 2014 στην τελευταία στήλη, αυτό τι μας δείχνει πρώτον, ότι οι αριθμοί των επιθεωρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά και το ποσοστό εκτός Ευρώπης επίσης. Εντός Ευρώπης είναι αυτό που βλέπετε με μοβ χρώμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι το μπέζ αμέσω μετά και το υπόλοιπο είναι έλεγχοι εκτός. Και το μισό περίπου των ελέγχων του 2014 ήταν εκτός Αμερικής και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Μέση Ανατολή, ε, Ειρηνικός, Ρωσία, Αφρική κτλ. Θα συνεχίσουμε ε, να διατηρούμε αυτούς τους ρυθμούς και Έδειξε η προηγούμενη διαφάνεια λοιπόν ότι υπάρχει διεθνής δραστηριότητα και υπάρχουν και στοιχεία των επιθεωρήσεων εξ ονόματος των κρατών μελών για να δίνουν τις άδειε. Από Ευρωπαίους επιθεωρητές αυξάνεται ο ρυθμός των επιθεωρήσεων. Έχουμε ε, όλο και περισσότερες συμβάσεις ε, με τους διεθνείς ε, ε, τους εκάστοτε εθνικούς οργανισμούς, Ινδία, Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ελέγχουμε μόνο τις κλινικές πρακτικές αλλά και τον τρόπο που παρασκευάζονται τα φάρμακα. Ε, έχουμε στοιχεία ε, για τα αποτελέσματα και έχουμε και εκπαίδευση. Οι πολλοί επιθεωρητές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιούνται πάρα πολύ σε κλινικές δοκιμές και ε, συμμετέχουν σε εκπαίδευση που διοργανώνουμε εμείς και οι εθνικές αρμόδιες ε, αρχές. Επίσης, παρακολουθούμε και τα αρνητικά αποτελέσματα ε, των ελέγχων και των επιθεωρήσεων την Αμερικανική Αρμόδια Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και άλλους διεθνείς φορείς. και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν αφαιρεθεί και άδειε για ε, κλινικές δοκιμές για βιοϊσοδυναμία αμερικανική πλευρά. Έχουμε στενή συνεργασία ιδιαίτερα με την FDA, την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, γιατί αν συντονίσουμε τις ε, δυνάμεις μα ε, μπορούμε να ελέγχουμε πάρα πολλές ε, δοκιμές και καλό είναι να μοιραζόμαστε αυτές τις προφορίες για να μην ελέγχουμε δύο φορές οι Αμερικανοί και εμείς, ε, να μην πολλαπλασιάζονται οι έλεγχοι, να πηγαίνουμε σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά κέντρα και να ανταλλάσσουμε όχι μόνο τα αρνητικά αλλά και τα θετικά στοιχεία και να τα ε, συμπεριλαμβάνουμε στον προγραμματισμό και το σχεδιασμό μας. Ε, κλινικές δοκιμές και μελέτες βιοϊσοδυναμίας για τα γενώσιμα σε συνεργασία ε, με την Αμερική από τον περασμένο Ιανουάριο, με κοινά ε, συστήματα ελέγχων, επιθεωρήσεων, κλινικών εργαστηρίων κτλ. Και συνεργαζόμαστε πολύ πιο στενά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να οικοδομήσουμε, θέλετε, ένα παγκόσμιο σύστημα, ένα κατάλογο των ε, εργαστηρίων, των δοκιμών, των αποτελεσμάτων και επαναλαμβάνω και τα θετικά και τα αρνητικά για να αυξηθούν οι προδιαγραφές και τα πρότυπα και σε διεθνές επίπεδο. Ήδη αναφέρθηκα στα θέματα της ε, εκπαίδευσης. Εμείς ε, ζητάμε από αρχές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινική Αμερική, Ρωσία, Αφρική να συμμετέχουν στα σεμινάρια μας και στα ετήσια εκπαιδευτικά μας προγράμματα για τους Ευρωπαίους εκπαίδευτες. Πέρυσι ξεκινήσαμε και ένα, μια εκπαίδευση κατάρτισης online σε συνεργασία με την Γαλλική Υπηρεσία Υγείας. Έχουν πράγματι ειδικέ εμπειρίες σε σχέση με την παρακολούθηση ε, της κατάρτισης των ελεγκτών σε συνεργασία και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ε, γιατί αυτές οι κλινικές τώρα έρευνες είναι βασικές. Ε, τα γενώσιμα είναι αντίγραφο του αρχικού φαρμάκου και αυτά τα γενώσιμα φάρμακα είναι σε θέση να κυκλοφορήσουν όταν λήξει η περίοδος αποκλειστικής χρήσης της ουσίας από την, για το πρωτότυπο φάρμακο. Υπάρχουν δύο-τρεις μελέτες α, οι οποίες γίνονται πριν κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο φάρμακο και υπάρχει διασταύρωση ε, των φακέλων από τις επιχειρήσεις. Αυτή η μελέτη της βιοϊσοτιμίας, να τη λέγαμε, είναι κάτι το οποίο ε, εμπλέκει 20, 24 η, η οι μελέτες, 24 οι υγιείς ασθενείς, ε, ε, οι οποίοι παίρνουν φυσικά και στις δοκιμές αυτές αντίστοιχες ποσότητες φαρμάκων πρωτοτύπων, γενοσύμων και ουδετέρων. Και φυσικά ελέγχεται ή γίνονται προσεκτικές αιματολογικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμής αυτής, των ελέγχων αυτών. Τώρα το ποιος κάνει αυτές τις μελέτες βιοϊσιδυναμίας υπάρχουν συγκεκριμένες ε, επιχειρήσεις, οι λεγόμενες CRO, Contract Research Organizations, ε, εκεί παίρνουν ε, τα συγκεκριμένα φάρμακα, κάνουν τις κλινικές δοκιμές, καταγράφουν τα αποτελέσματα και επίσης γίνονται μελέτες μέτρησης της περιεκτικότητας των συγκεκριμένων φαρμάκων από εργαστήρια. Ε, λόγω του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εμπορία και η πώληση των συγκεκριμένων γενοσύμων ε, μπορεί να χρησιμοποιούνται πολλά ονόματα και πολλές επιχειρήσεις αλλά χρησιμοποιούν την ίδια ουσία, το ίδιο φάρμακο και τα ίδια πιστοποιητικά ε, βιοαντιστήχησης ή βιοϊσοδυναμίας. Πολλές εταιρείες λοιπόν μπορεί να τα εμπορεύονται αλλά βασίζονται στην ίδια μελέτη και γι' αυτό οι μελέτες αυτές λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Α, ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν αδειοδότηση από τις ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας Προσπαθούμε εμείς να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες θεωρούμε ότι απαιτείται να υπάρξουν επιθεωρήσεις ανάλογα με την ιστορία ε, της συγκεκριμένης εγκατάστασης και επιχείρησης. Mm. Αν δεν υπάρχει στο παρελθόν έλεγχος αυτό είναι ένας παράγων ο οποίος μας οδηγεί στην ε, ε, διοργάνωση ενός ελέγχου και ελέγχουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι κλινικές αυτές δοκιμές, ε, ε, τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι αιματολογικές εξετάσεις κτλ. Η ευθύνη για τις δοκιμές αυτές γίνονται φυσικά, ή μάλλον έγκυται η ευθύνη σε αυτόν ο οποίος χρηματοδοτεί την κλινική δοκιμή. Είναι υπεύθυνο επίσης και για την ποιότητα των δεδομένων και στο τέλος αυτός είναι ε, ο υπεύθυνος για να πωλήσει το συγκεκριμένο φάρμακο στους ε, Ευρωπαίους διανομής. Συνεργάζονται τα κράτη-μέλη και το EMA ε, εδώ και χρόνια στην διεξαγωγή ενός ελέγχου ετησίου, ενός προγράμματος ετησίων ελέγχων αυτών των οργανώσεων οι οποίες λειτουργούν υπεργολαβικά, των CRO. Εδώ θα δείτε ότι αντίθετα με την κατανομή των δοκιμών των καινοτόμων, εδώ μιλάμε στις μελέτες οι οποίες έχουν κάνει σε επίπεδο βιοδυναμίας, στις χώρες όπου γίνονται οι έλεγχοι είναι στην Ινδία, 105 συνολικά 143 μαζί με τα καινοτόμα προϊόντα, Ιταλία, Καναδάς, Ρωμανία και Γερμανία. Στην Γερμανία βλέπετε ότι αντίθετα με την Ινδία είχαμε χίλιες επιθεωρήσεις, μόνο 19 από αυτές αφορούν γενώσιμα. Οι άλλες κλινικές δοκιμές αφορούν νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ δραστήριο πρόγραμμα ελέγχου και όπως βλέπετε στην Ινδία 105 μετά από διαδικασίες αδειοδότησης σε εθνικό επίπεδο. Το GVK Bioscience είναι μία από αυτές τις επιχειρήσεις. Ε, η Γαλλική Υπηρεσία έκανε εννέα δοκιμές τις οποίες διεξήγαγε η εταιρεία GVK Biosciences έδειξε ότι στο τέλος υπήρχαν κάποια προβλήματα με κάποιες μελέτες ηλεκτροκαρδιογραφημάτων αλλά κατά τα άλλα ε, τα ECGs από την ίδια μελέτη είχαν ε, επισημανθεί με διαφορετικά ονόματα Ίσως ε, εδώ μπορεί κανείς να δώσει πολλές εξηγήσεις, δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί υπήρξαν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αυτές οι παραβάσεις έγιναν από το 2008 μέχρι το 2014 και αφορούσαν πολύ προσωπικό ε, των κλινικών ε, της GVK Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δοκιμές αυτές και η εμπιστοσύνη στο ποιοτικό σύστημα της κλινικής αυτής του GCP είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί η εμπιστοσύνη έχει μειωθεί. Ε, γίνεται μια έγινε μια παράλληλη αγγλική έρευνα του εργαστηρίου αυτή τη φορά της GVK Biosciences αλλά δεν έδειξε να υπάρχουν συστηματικά προβλήματα ή τουλάχιστον προβλήματα τα οποία να παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν μετά από τις πληροφορίες τις οποίες πήρε από τη Γαλλική Υπηρεσία επί τη βάση του άρθρου 31 της Οδηγίας 83-2001 που ασχολείται με το θέμα αυτό, που καλύπτει το θέμα αυτό, αποφάσισε να ελέγξει τις μελέτες τις οποίες έκανε η GVK και πριν από το 2008 και τα ευρήματα υπονομεύουν την αξιοπιστία των δοκιμών τις οποίες έχει κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία GVK και όλες ε, οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας της συγκεκριμένης εταιρείας GVK θεωρούνται αναξιόπιστες. Έχουμε λοιπόν τώρα το σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ευρήματα των δοκιμών αυτών και να τα αξιολογήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο CHMP και να μπορέσουμε έτσι να αναλάβουμε προληπτική δράση, ισχυρή δράση προστασίας των Ευρωπαίων ασθενών και αξιολόγησης επαρκούς και αποτελεσματικής των, ε, δοκιμών βιοϊσοδυναμίας. Ε, οι δοκιμές αυτές πολλές φορές όπως είπα αφορούν πάρα πολλές επιχειρήσεις αλλά οι μεγάλες ε, επαγγελματικές ε, κλινικές μπορεί να κάνουν 150 τέτοιες δοκιμές σε αιτήσια βάση. Όταν βλέπουμε μία περίοδο δεκαετίας βλέπουμε φυσικά ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ υψηλός. Για 300 από αυτές τις δοκιμές υπήρξαν και από άλλες πηγές επαρκή υποστηρικτικά στοιχεία για την αξιοπιστία τους και παραμένουν στην αγορά της Ευρώπης. Αλλά για φάρμακα τα οποία δεν έχουν από άλλες πιο σίγουρες πηγές δεδομένα τότε το CHMP σύστησε την διακοπή διανομής των φαρμάκων αυτών εκτός και αν είναι κρίσιμης σημασίας για τους ασθενείς γιατί δεν θα υπάρξουν εναλλακτικά φάρμακα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Ε, μπορεί να μην υπάρχουν λοιπόν για κάποιους ασθενείς εναλλακτικές φαρμακευτικές ουσίες και γι' αυτό θα συνεχίσουν να παίρνουν τα συγκεκριμένα φάρμακα αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν νέες μελέτες βιοϊσοδυναμίας στους επόμενους 12 μήνες και να υποβάλουν επιμέρους στοιχεία. Λοιπόν τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ε, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα μελλοντικά βήματα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η περίοδος αυτή ε, και ο τρόπος με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν τα CRO στις υπεργολαβικές αυτές κλινικές που κάνουν τις δοκιμές βιοϊσοδυναμίας ε, γιατί όπως είπα πολλές κάνουν ταυτόχρονα 30-40 τέτοιες μελέτες. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση ε, και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με τους διεθνείς εταίρους μας. Να φτιάξουμε ένα κοινό κατάλογο των ευρημάτων της αξιολόγησης των δοκιμών αυτών. Να υπάρξει υπεραιτέρω αύξηση σε διεθνούς ενημέρωσης γύρω από τα CROs σχετικά με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επιθεωρήσεων θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ε, ε, θα συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των μελετών τις οποίες περιλαμβάνουν στους φακέλους που υποβάλλουν για έγκριση οι, ε, οι, οι αυτές. Και τέλος θα περάσουμε στην εφαρμογή ε, της ε, σωστής ε, κατανομής των στοιχείων ενημέρωσης και των εμπειριών τις οποίες έχουμε, καλύτερο συντονισμός δηλαδή των ελέγχων τύπου GCP, όπως προβλέπεται από το νέο κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές γύρω από το πλαίσιο των γενοσύμων φαρμάκων όπως επίσης και γύρω από τις υπηρεσίες και τις κλινικές οι οποίες θα διασφαλίσουν νομίζω μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία στις επιθεωρήσεις αυτές. Αυτά. Merci, merci beaucoup, Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Σουίνι. Ο Ματίας Κρότε έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι. Βεβαίω, Είμαι ο σύνδεσμος του Κοινοβουλίου με τον ΕΟΦ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον κύριο Σουίνι, ε, για την παρουσίαση και την ερώτηση του κυρίου Λίζε, του εισηγητού. Ένα, ε, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ήταν χίλιες αιτήσει, χίλιες ε, υποθέσεις που έπρεπε να ε, επεξεργαστούν σε πολύ λίγο χρόνο το σύστημα λειτουργεί. Αλλά στο τέλος είπε ξανά ο κύριος Σουίνι και είναι τα διδάγματα που θα πρέπει να εξαγάγουμε για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, να συνεργαστούμε και με τους Αμερικανούς και με άλλους. Να μην πάμε να κάνουμε διπλούς και τριπλούς ελέγχους κάθε φορά. Διεθνώς να συντονιστούμε καλύτερα για να είναι το ε, δίχτυ πιο σφιχτό και πιο μικρά τα μάτια. Εγώ είμαι λίγο καιρό σύνδεσμος με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Έχω επικρίνει ότι δεν ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Βελτιωθήκατε. Λειτουργεί καλά τώρα το σύστημα και με ευχαριστώ γι' αυτό. Διαπιστώνουμε ότι αντιδράσατε ε, εγώ τα έμαθα από την τηλεόραση βασικά, από τις ειδήσει, φαντάζομαι και οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά κάπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σφίξουμε το δίχτυ ε, και διεθνώς. Διαπληκτιζόμαστε πολύ, συζητούμε για τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί τα συζητάτε, γιατί μόνο αρνητικά ακούμε για το TTIP. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε καλύτερα για διεθνείς ελέγχους και επιθεωρήσεις γιατί κλινικές δοκιμές οι μελέτες γίνονται σχεδόν αποκλειστικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι γίνεται με την ασφάλεια των αποτελεσμάτων. Και χωρίς συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εμείς μπορούμε να ασκήσουμε καμία πίεση έτσι ώστε τα πρότυπα των επιθεωρήσεων να αυξηθούν μαζί με τους Αμερικανούς, επαναλαμβάνω για την ασφάλεια. Περιμένω. Είμαι πολύ περίεργος. Ξέρω ότι δεν έχει αυτό το θέμα να κάνει με το συγκεκριμένο, αλλά το TTIP το συζητήσαμε αυτή την εβδομάδα και όχι μόνο εδώ και σε όλο το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και πάλι. Πολύ γρήγορα αντιδράσατε. Μπράβο σας. Και αξίζεται πολλά συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο έπαινο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρότ. Τώρα ο κύριος Μπιούτσα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πάρα πολύ πλήρης η παρουσίαση. Ακούσαμε τις δύο παρουσιάσεις που περίχαν τόσες πληροφορίες αλλά με ανησύχησαν μερικά. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης εκεί δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί υπάρχουν κανονισμοί, λομικές λύσεις και αφορούν και τα, τη φαρμακοβιομηχανία και τις κλινικές δοκιμές. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και υπάρχει απ' την άλλη το θέμα των τρίτων χωρών που μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο μέρη. Τις Ηνωμένε Πολιτείες όπου η FDA από ό,τι ξέρω διαφέρει από την αίμα στις διαδικασίες της. Άρα πού βρισκόμαστε ως προς το συνδυασμό, ως προς την συγκρισιμότητα των προτύπων μας και εκείνων. Και υπάρχει η όχι αμοιβαία αναγνώριση των αμερικανικών φαρμάκων από την αίμα και το αντίστοιχο, το αντίστροφο. Μπορεί να υπάρχουν σκάνδαλα στην ε, γραφή και αδειοδότηση ορισμένων φαρμάκων και που να καταλήγουν σε αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι το πρώτο μετά οι άλλες τρίτες χώρες που είναι οι αναπτυσσόμενες Ινδία, Πακιστάν, Κίνα. Εδώ με ανησυχεί κάτι. Δεν υπάρχει αρκετό συντονισμός. Το θέμα είναι απλό. Η λήψη φαρμάκων. Το, η ενεργός ουσία είναι η ίδια παντού. Υπάρχουν βέβαια πολλές ουσίες και φάρμακα, αλλά δεν πρέπει κανονικά να υπάρχει πρόβλημα αφού η ενεργή ουσία έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια υπηρεσία. Η δραστική ουσία μάλιστα θα έλεγα. Επομένως έχει γίνει έλεγχος και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε ίσως να διαπιστώσουμε αν όντως έχει γίνει αλλά τέλος πάντων το πρόβλημα που θέτω είναι το εξής η ΕΜΑ έχει εμπιστοσύνη στις μονάδες που κάνουν αυτές, αυτούς τους ελέγχους. Υπάρχει κανένα είδος πιστοποίησης, αδειοδότης, κάτι που να δείχνει, να αποδεικνύει τι έχει γίνει στις δοκιμές. Θα ήθελα να το ξέρω αυτό γιατί με ενδιαφέρει και για τα γενώσιμα φάρμακα αλλά και για τα καινούρια φάρμακα που είναι πολύ σημαντικά για τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχουν οι τεράστιες αυτές εταιρείε και άρα πρέπει και η Ένωση να παίξει κάποιο ρόλο. Πολλές φορές οι κλινικές αυτές δοκιμές των καινούργιων φαρμάκων γίνονται σε τρίτες χώρες λόγω του ότι πιο εύκολα πείθεται ο κόσμος να τα δοκιμάσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, ε, ΕΟΦ για την τεράστια προσπάθεια την οποία έχουν κάνει και για τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Συμμερίζομαι πλήρως αυτά τα οποία είπε ο Πέτερ Λίζε για την ε, υποτιθέμενη απουσία κινδύνων στις κλινικές δοκιμές. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. με ενοχλεί επίσης και η κοινωνική διάσταση αυτών των δοκιμών που γίνεται σε πληθυσμούς οι οποίοι είναι κοινωνικά ευάλωτοι. Τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό ε, των ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών ε, έγιναν τέτοιες δοκιμές και με παιδιά τα οποία δεν ήξεραν τι ουσίες έπαιρναν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εις βάρος των φαρμακευτικών ε, ε, εταιριών οι οποίες έχουν κάνει αυτές τις κλινικές δοκιμές ακόμα και αυτές που προηγούνται των κλινικών δοκιμών κατεξοχήν. Πώς μπορούμε λοιπόν να οργανώσουμε τους ελέγχους αυτούς σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, όχι μόνο με τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και με τις τρίτες χώρες τις οποίες δεν υπάρχει ε, επαρκής έλεγχος για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δεν ξέρω κύριε Λίζε αν θέλετε ξανά το λόγο. Όχι. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Ις, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ρίς λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Καταρχάς σε διεθνές επίπεδο συνεργαζόμαστε με την Αμερικανική ε, Υπηρεσία, την ομόλογή μας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πράγματι ένα σύστημα που θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις χώρες τις οποίες θα πρέπει να ελέγχουμε περισσότερο όπως την Κίνα, την Ινδία κτλ. οι συζητήσεις του TIP, του TTIP ε, μας δίνουν μια αφορμή επιπλέον για να ελέγξουμε λίγο αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε και τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να το πετύχουμε. Σχετικά τώρα με τη διεθνή κοινότητα υπάρχει δυνατότητα οργανωμένων συναντήσεων των ε, ε, αρχών εποπτείας από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, η Βραζιλία, η Νότια Κορέα, που ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία κάνουμε και θέλουν να τα κάνουμε όλοι μαζί καλύτερα. Μεταρρυθμίζουμε επίσης ε, και την Διεθνή Διάσκεψη ε, Εναρμόνισης που είναι η νομική διαδικασία την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε ε, για να υπάρξει σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνώριση δοκιμών, φαρμάκων κτλ. Άλλες χώρες βέβαια είναι πολύ δραστήριες, άλλες είναι λιγότερο δραστήριες. Σχετικά τώρα με τον αριθμό των κλινικών δοκιμών για τα παιδιά, από η απάντησή μας είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει ο σωστός έλεγχος των επιθεωρήσεων έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, ε, τέτοιου είδους ε, δόκιμες ακόμα και για παιδιά αν αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείες κυρίως. Θα πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι ανεξαρτήτως της φύσης αυτών των δοκιμών ελέγχουμε πάντα και φροντίζουμε και όταν δεν αρκεί το GCP τότε προφανώς και οι έλεγχοι του GCP θα πρέπει να εφαρμόζονται περαιτέρω έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ δόκτωρα. αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις τις συγκεκριμένες ο, ο Αναφέρθηκε επίσης ε, και στο θέμα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων και στις σχέσεις ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές ε, και στη σχέση ανάμεσα στις αμερικανικές υπηρεσίες ε, και τις δικές μας υπηρεσίες με τις ομάδες κλινικών δοκιμών και τα GRPs είμαστε σε ε, συνεχή επαφή, εβδομαδιαία επαφή με τηλεδιασκέψεις, με αμοιβέ ενημερώσεις. Μπορούμε να αναλάβουμε λοιπόν κοινή δράση στα πλαίσια των GCP και ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιούμε και τις εταιρείε τις οποίες έχουν ελέγξει οι Αμερικανοί και τα αποτελέσματα είναι θετικά και ελέγχουμε άλλες εταιρείες, έτσι δημιουργείται μια θα έλεγα συνεργατική σχέση με τις αμερικανικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα και οι καρποί αυτών των κλινικών δοκιμών είναι για την Ευρώπη και για τους Αμερικανούς ωφέλιμα και χρήσιμα και ε, υπακούν σε συγκεκριμένα επίπεδα Νομίζω ότι ακόμα και αν διαφέρουμε σε επίπεδο μεθοδολογίας η ουσία είναι μία και για τις δύο ε, περιοχές. Απαιτείται η ίδια περίπου χρονική διάρκεια, απαιτείται η ίδια διαδικασία δημιουργίας ε, οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης και αν τυχόν υπογραμμίσουν κάπου ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα δράσουμε από κοινού για να το αντιμετωπίσουμε. Προβλήματα υπάρχουν, έχουμε βρει τέτοια προβλήματα, έχουμε συνεργαστεί στους ελέγχους σαν παράδειγμα κάποιων κλινικών και με τον Διεθνή Οργανισμό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος μας είναι να βάλουμε σε ένα κατάλογο όλες αυτές τις ε, επιχειρήσεις και για την προστασία των ε, συμμετεχόντων, των ευάλωτων αυτών κοινωνικών κατηγοριών. Ε, οι επιθεωρητές και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ε, επίσης δημοσιεύσει συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας των συμμετεχόντων στις κλινικές αυτές δοκιμές και αυτό φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους επιθεωρητές. Πάντως ε, οι επιθεωρητές συμμετέχουν όλο και περισσότερο στις δοκιμές αυτές που γίνονται σε τρίτες χώρες και η νομοθεσία στην Ινδία σχετικά με τις κλινικές δοκιμές έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια για την προστασία, την καλύτερη προστασία των ευάλωτων πολιτών που συμμετέχουν σε αυτές τις κλινικές δοκιμές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και για την ποιότητα της συζήτησης πάρα πολύ σημαντική. Και τώρα ένα τρία θέματα. Οι συνάδελφοι στις τοποθετήσεις ε, θέλησαν να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να εντείνουν τους ελέγχους. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός αυτός στις 16 Ιουνίου του 2014 θα πρέπει να ε, καταγράφονται οι κλινικές δοκιμές, ε, αλλά ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ μόνο στις 28 Μαΐου του 2016 ουσιαστικά. Και ε, θα πρέπει πραγματικά οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Αυτή τη στιγμή σε τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Στο 21 διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. για την εργασία τους. Ε, την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα είναι στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2015. Καλώς σας βράδυ.